Γεια σας. Καλώς ήρθατε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Αν και είμαστε σε μικρό αριθμό ακόμη, είμαστε μόνο δύο-τρεις όλοι και όλοι, ας περιμένουμε λίγα λεπτά για να μπορούμε να αρχίσουμε με περισσότερα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας. Το πρώτο μας ε, θέμα θα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών. Σε λίγα λεπτά. The representatives of the energy community. Uh, dear colleagues, uh, uh, Περιμένουμε λίγα λεπτά. dear friends. Περιμέναμε 10 λεπτά το φίλο μας τον κύριο Κόχλιτσεκ. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Προτεραιότητες της Επιτροπής μας στον προϋπολισμό το 2018, ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εισηγητής του προϋπολογισμού είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε που ήρθατε. Να αρχίσουμε λοιπόν με δική σας πρώτη βασική τοποθέτηση. Είναι βέβαια μεγάλη σημασία του ετήσιου προϋπολογισμού για την επίτευξη των προτεραιοτήτων στους τομείς πολιτικής της Ένωσης. Και υπενθυμίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού 2018 τα τέλη, μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ανάμεσα στη δημοσίευση του σχεδίου και της ψήφου του προϋπολογισμού στις 20 Ιουνίου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών λοιπόν θα ψηφίσει μόλις ένα μήνα μετά. Πρέπει η γνωμοδότησή μας να λάβει τη μορφή επιστολής γιατί δεν είναι διαφορετικό, διαφορετικά δυνατό να προλάβουμε, δηλαδή να εκδώσουμε γνωμοδότηση με συμβαστικές τροπολογίες κλπ. Δεν έχουμε χρόνο. Άρα στην βάση των τρεχουσών συζητήσεων ιδίως ο συναδελφός μας Ζίκφριτ Μόρεσον και ε, βάσει τις προτάσεις του Ζίκφριτ Μόρεσον και στα σχόλιά του με βάση αυτά θα στείλω επιστολή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η ψήφος σχεδιάζεται να γίνει εδώ στις 11 Εβδόμου και στις 25 Σεπτεμβρίου του 2017 θα ψηφιστεί το ψήφισμα για τον προϋπολογισμό. για να προλάβουν να ληφθούν υπόψη οι απόψει της Επιτροπής Ήτρε. Μπορείτε να τοποθετηθείτε για θέματα πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων εφόσον τα στείλετε μέχρι τις 27 Απριλίου στη γραμματεία της Επιτροπής Ήτρε, δηλαδή σε δύο-τρεις ημέρες. Δυστυχώς είναι πολύ σύντομο το χρονικό αυτό διάστημα. Αλλά καλείστε να υποβάλλετε ιδέες για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις για του χρόνου, 2018, του, του παραχρόνου δηλαδή, μέχρι 27 Απριλίου. Να παρακαλέσουμε τώρα τον συνάδελφό μας τη επιτροπή Προπολογισμών να τοποθετηθεί πρώτος στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσά αγαπητοί συνάδελφοι που με καλέσατε σήμερα και με δέχεστε εδώ για να συζητήσουμε για τι προτεραιότητε του, προπολογισμού της Ένωσης. Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο εγκρίθηκε η έκθεσή μου για τις βασικές κατευθύνσεις του προπολογισμού του επόμενου χρόνου και σε αυτές τις βάσεις το Κοινοβούλιο τοποθετεί τις πολιτικές προτεραιότητες που θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον νοσιακό προϋπολογισμό του χρόνου. Το επόμενο βήμα είναι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέλη Μαΐου και μετά θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα ήθελα τώρα να συζητήσω πρώτα μαζί σας τις πολιτικές προτεραιότητες όπως τις υποβάλλω εγώ στην έκθεση που όπως είπα εγκρίθηκε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Πιο πολύ όμως με ενδιαφέρει να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με τα σημεία που θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και ε, απέναντι στην Επιτροπή και απέναντι στο Συμβούλιο. Ποιο το μπει, δηλαδή θα πρέπει να επιμείνουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν στους επόμενους μήνες. Εγώ έχω προωθήσει δύο σημαντικέ πολιτικέ προτεραιότητε Ανάπτυξη και εργασίε, δουλειέ και δεύτερο ασφάλεια των πολιτών γιατί νομίζω ότι αυτά χρειάζονται οι ε, πολίτες της Ευρώπης, δηλαδή δουλειές και ασφάλεια. Για το πρώτο και την πρώτη προτεραιότητα, ανάπτυξη και δουλειές. Νομίζω ότι η Επιτροπή σας έχει κέριο ρόλο να παίξει. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη και απασχόληση και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τον προπολογισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε και να κάνουμε πιο ανταγωνιστική την οικονομία μας και για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται καινοτομία έρευνα, υποδομές. Αυτά είναι βασικά στοιχεία και στους τομείς αυτούς ηγείται η Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να ενισχυθούν ο Horizon 2020, η ε, ε, διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, το κόσμε, ο έρασμος και βεβαίως η πρωτοβουλία εγγύησης για την νεολαία, διότι οι νέοι αξίζουν την υποστήριξή μας. Άρα λοιπόν τα προγράμματα που προανέφερα, όπως COSME 2020 κλπ. πρέπει να ενισχυθούν και για τον ορίζοντα 2020 πιο συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός εγκρίσεως σχεδίων, project, υπό τούτο εδώ το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ πιο ισχνός από ό,τι πριν. Είναι 20% τώρα. Ήταν Τώρα είναι μόνο 13%. Δηλαδή έχουμε επιτύχει να χρηματοδοτήσουμε μόνο 13%. Ενώ στο προηγούμενο ΠΔΠ ήταν 19%. Άρα έχει μειωθεί ο ρυθμός για δύο λόγους. Πρώτον, λαμβάνουμε πολλές αιτήσει που καμιά από αυτές δεν ε, οι πολύ λίγες είναι καλές. Δεύτερον, υπάρχουν λιγότερα κονδύλια. Είναι περισμένα τα κονδύλια μας για τον 2020 και επηρεάζονται και από τη δημιουργία του EFSI επειδή εγώ θέλω να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καλά έργα, καλά project που ζητούν χρηματοδότηση, είναι καλό που υποβάλλονται πολλές αιτήσει. Θα χρειαστεί λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του ορίζοντος 2020, ο οποίος υπέστη τις επιπτώσεις του EFSI που ήταν σωστό να γίνει το EFSI, το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων, για να κλείσουν τα κενά επενδύσεων. Ορισμένες από τις επιπτώσεις θα έρθουν με την αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και θα προσθεθούν 200 εκατομμύρια όταν θα εγκριθεί η αναθεώρηση. Αυτό είναι καλό σημάδι. Ήθελα επίσης στον προπολογισμό του επομένου έτους να αυξηθούν οι πιστώσεις ιδίως για προγράμματα βασικής έρευνας όπως το πρόγραμμα Marie Curie και το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Όπως είπα λοιπόν, καινοτομία, έρευνα, πρώτη σημαντική προτεραιότητα. Υποδομές επίσης, διότι ενισχύουν την οικονομία, την κάνουν πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική προς τους επενδυτές, ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί απασχόληση, ε, διευκόλυνση στην Ευρώπη, κόσμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση τη νεολαίας και βεβαίως το πρόγραμμα Έρασμος. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ως κοινοβούλιο έχουμε παίξει τον ρόλο μας. Σας ενημερώνω θα πρέπει να το γνωρίζετε, διότι όπως είπα έχουμε παίξει τον ρόλο μας και τώρα ο φάκελος έχει τεθεί υπόψη του Συμβουλίου. Υποτίθεται ότι θα τεθεί υπόψη σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και δεν θέλουν να εγκριθεί η αναθεώρηση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ πριν από τις εκλογές που θα γίνουν στις 8 Ιουνίου στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν έχει άμεση επίπτωση. Θα υπάρξει εάν δεν εγκριθεί η αναθεώρηση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Διότι αυτή επιτρέπει να επαναδιατεθούν 200 εκατομμύρια, 100 για τον έρασμο και 100 για το πρόγραμμα COSME. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αν δεν εγκριθεί αμέσως εάν καθυστερήσει έστω και για πολλούς μήνες. Θα υπάρξει όμως σοβαρός κίνδυνος για project τα οποία είναι σημαντικά και για τη δική σας επιτροπή αλλά που και για μένα αποτελούν πολιτική προτεραιότητα εάν τελικώς δεν εγκριθεί η αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου καθόλου. Τώρα, για το FC2. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το FC2, πρότειναν περιορισμένο επανακαθορισμό για ορισμένα ε, κονδύλια του ΣΕΦ. Εμείς είπαμε όχι, διότι επηρεάζονται από την δημιουργία του FC1 και οι εισηγητές του FC2 προτείνουν να μην γίνουν άλλες περικοπές στα χρήματα της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη, θεωρούν ότι όλα τα χρήματα για το FC2 θα πρέπει να είναι νοπό χρήμα. Αυτή είναι και η δική μου θέση και γνώμη. Στις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού του επομένου έτους θα υποστηρίξουμε μια θέση που θεωρούμε ότι απηχεί τα συμφέροντα και της Επιτροπής ΙΤΕ, δηλαδή να μην περικοπούν τα κονδύλια της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη όταν θα εγκριθεί το FC2. Πιο συγκεκριμένα για την Επιτροπή σας, πέρσι, στην διαδικασία του προπολογισμού, το Συμβούλιο πρότεινε την περικοπή κάποιων διοικητικών δαπανών οργανισμών που έχουν σχέση με την εφαρμογή του οριζόντος 2020 και ορισμένων κοινοπραξιών. Εμείς ως κοινοβούλιο είπαμε όχι και επαναφέραμε τους αρχικούς αριθμούς της Κομισιόν. Αυτή θα είναι και η δική μου θέση τώρα. Με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να δεχθώ μείωση των διοικητικών δαπανών οργανισμών οι οποίοι εργάζονται για τον ορίζοντα 2020 και για κοινοπραξίες ε, ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Υπάρχει ένας οργανισμός Οργανισμός Συνεργασίας για την Ενεργειακή Ένωση που ζήτησε το προσωπικό της να αυξηθεί κατά 30 οργανικές θέσεις γιατί έχουν αναλάβει νέα καθήκοντα. Μετά από την ενημέρωση της νομοθεσίας για την ασφάλεια προμήθειας αερίου και γιατί μπαίνουν σε νέους κώδικες κλπ. Ζήτησαν λοιπόν ο προϋπολογισμός τους να φτάσει τα 19,95 εκατομμύρια ευρώ αντί των 13 που είχε προβληθεί για φέτος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει νόημα. Είναι λογικό, διότι έχουν αναλάβει περαιτέρω καθήκοντα. Θα ήθελα όμως να γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη της δικής σας Επιτροπής επ' αυτού. Και αν θα πρέπει όντως να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Συνεργασίας για την Ενεργειακή Ένωση. Και αν αυτό θα περιληφθεί στην επιστολή που πρόκειται να μας απευθύνεται στο όνομα της Επιτροπής σας, Επιτροπής Ήτρε. Θα είναι πολύ χρήσιμο, εάν δηλαδή, να γνωρίζουμε, εάν δηλαδή η αίτηση είναι θεμελιωμένη για αύξηση της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι εσείς είστε περισσότερο σε θέση να γνωρίζετε εάν αυτό είναι δικαιολογημένο. Τέλος, πιλωτικά προγράμματα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές. Όπως γνωρίζετε υπάρχει προϋπολογισμός για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα προχωρήσουμε σε εξή. Θα προτείνουμε ένα πακέτο πιλωτικών προγραμμάτων που θα τα προτείνουμε για χρηματοδότηση στη βάση προτάσεων που θα προέρχονται από διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Θα προχωρήσουμε ακριβώς όπως πέρσι. Θα είμαστε εις θέση να περιλάβουμε προ χρηματοδότηση μόνο πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προαξιολόγηση και έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια βαθμολόγηση α ή β. Πιλωτικά προγράμματα που λαμβάνουν βαθμό γ ή και χαμηλότερο, όπου δηλαδή θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι καλά, δεν θα μπορέσουν να περιληφθούν στο πακέτο χρηματοδότησης. Όσα λάβουν βαθμολόγηση α έχουν πολλές πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν, και πιθανότητες να χρηματοδοτούν έχουν και τα Β. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις σας είναι σημαντικό να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προαξιολόγηση. Προθεσμία υποβολής project στην Κομισιόν είναι η 3η Μαΐου, 3η Πέμπτου. Οποιοδήποτε πιλωτικό πρόγραμμα ή προπαρασκευαστική δράση που επιθυμείτε να υποβάλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβαστεί σε αυτήν μέχρι την 3η Μαΐου. Νομίζω ο πρόεδρος σας είπε ότι θα πρέπει να διαποβάλλετε πρώτα στη γραμματεία της Επιτροπής σας. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτό. Ο πρόεδρος γνωρίζει καλύτερα τις λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η τελική καταληκτική ημερομηνία που θα πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 3η Μαΐου, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα αξιολογήσει και εν τέλει θα γνωρίζουμε ποια είναι η γνώμη της, εάν ναι ή όχι θα πρέπει να περιληφθούν στο τελικό φάκελο. Εγώ θέλω να δώσω στο δυνατόν περισσότερα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστική δράση. Εμένα βέβαια τη, τη δουλειά μου θα την κάνετε πιο δύσκολη γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε περισσότερη επιλογή. Αλλά θέλω να κατατεθούν καλά πιλωτικά προγράμματα, να έχουμε ένα μεγάλο εύρο τέτοιων προγραμμάτων για να μπορέσουμε να επιλέξουμε, έστω και αν δυσκολευτεί το έργο μου γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε επιλογέ. Σα ενθαρρύνω όμω να υποβάλλετε, να καταθέσετε οποιαδήποτε πιλωτικά προγράμματα ή προπαρασκευαστικέ δράσει που ενδέχεται να έχετε στο μυαλό σα θεωρώ ότι η σημερινή συνάντησή μα θα αποτελέσει την αφετηρία τη συνεργασία μα. Είναι πολύ σημαντικό όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο προπολογισμού στα τέλη Μαΐου και θα βάλει τα νούμερα στο τραπέζι να παραμείνουμε σε επαφή. Να βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο διότι οι προτεραιότητές σας συμπεριλαμβάνονται και στις δικές μου. Δηλαδή καινοτομία, έρευνα, υποδομές από τη δική μου πλευρά λοιπόν η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή. Ελπίζω η σημερινή λοιπόν συνάντησή μας να αποτελέσει την αφετηρία και όχι το τέλος της συνεργασίας μας. Πρόεδρο. πράγματι, πολύ σημαντικέ συζητήσει αυτές για τον προϋπολογισμό του 2018 βεβαίω έτσι. Δεν θα έχουμε πολλέ δυνατότητε. Το πιο σημαντικό θα είναι η επιστολή που θα στείλω στην Επιτροπή Προπολογισμών και βεβαίω θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο πριν από το ψήφισμά μα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Πρώτα όμω προηγείται η σημερινή μα συζήτηση, αυτή που διεξάγεται τώρα ιδέες για ε, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Ο συνάδελφός μας της Επιτροπής Προϋπολογισμών επανέλαβε αυτό που είπα και εγώ στην αρχή. Είναι σημαντικό λοιπόν να υποβάλλετε τέτοιες ιδέες στη γραμματεία μας μέχρι 27 Απριλίου. Τρεις μέρες σας μένουν ακόμη. Λιγότερο από τρεις. Ευχαριστώ. Τώρα, επειδή αισθάνομαι και υπεύθυνο ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Ήτρε επτά θέματα. Πρώτο, πρώτο λοιπόν, γνωρίζουμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο. Πρώτο λοιπόν. Δεύτερο, ευχαριστώ πολύ που στοχεύετε, που εστιάζετε τόσο πολύ στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Τρίτο, Εμείς που αισθανόμαστε και υπεύθυνοι για την πραγματική οικονομία, γεωργία βεβαίως, και αυτό είναι ε, πραγματική οικονομία, δεν υπάρχει εμφωλία και η γεωργία. Όμως όλα τα υπόλοιπα, ίσως ορισμένα να υπάγονται σε αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πάντως η πραγματική οικονομία είναι εδώ, στη δική μας Επιτροπή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε, να σεβόμαστε τις ε, υφιστάμενες δεσμεύσεις, υποσχέσεις, διότι η πραγματική οικονομία δεν δέχεται αλλαγές στη χρηματοδοτική μας υποστήριξη. Τέταρτο, είναι πολύ σημαντικό να αποφευθούν περικοπές σε υφιστάμενα προγράμματα που τρέχουν ήδη. Πέμπτο, αυτό θα είναι κάπως μακροσκελέστερο, διότι καθορίσατε την προσέγγισή σας στα δημοσιονομικά θέματα με γενικούς όρους. Έχετε δίκιο ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τους πολίτες και η εξωτερική και από την σκοπιά αυτή έχουμε κάποιες υποχρώσεις. Για παράδειγμα, ασφάλεια παροχής ενέργειας, που και αυτό είναι δική μας ευθύνη και μπορεί να διασυνδεθεί μάλιστα και με τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Σημαντικό αυτό και συνεργασία μας με την Ενεργειακή Ένωση. Αν και δεν είναι τόσο πολύ αυτό στόχευση της δικής μας Επιτροπής. Όμως περισσότερο είναι η εσωτερική ασφάλεια. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, κυβερνοασφάλεια. Μερικά άλλα πράγματα. Ας τα λάβουμε λοιπόν, υπό, λοιπόν υπόψη. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι η κοινωνική ασφάλεια αν μιλούμε για εξωτερική, εσωτερική και κοινωνική ασφάλεια, θεωρούμε ότι είμαστε απολύτως υπεύθυνοι, διότι η Επιτροπή Απασχολήσεω, πολύ σημαντική για μας, μπορεί και αυτή να δραστηριοποιείται εφόσον εμείς δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, βιομηχανία και Φθήνη ενέργεια, χαμηλέ τιμέ, ασφάλεια τη προμήθεια ενέργεια κλπ. Το είναι το πιο σημαντικό. Καινοτομία έρευνα. Ασφαλώς και είμαστε υπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν στον χώρο αυτό. Χρήματα για το EFSI γνωρίζουμε επίσης ότι για την καινοτομία και έρευνα. Δεν πρόκειται μονάχα για ένα, δύο ή τρία έτη και τα αποτελέσματα αυτών των ετών. Πρόκειται για μακροπρόθεσμη προοπτική. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς όμως ότι θα πάψει η επιρροή στην οικονομία μας μέσα σε 5 ή 10 χρόνια. Άρα μην ανακόψετε ή τέλος πάντων θα πρέπει να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε περικοπή στα ε, προγράμματά μας. Το πρόγραμμα Μαρή Curie Σκοντόφσκα για την νεολαία, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε τέτοια Μάλιστα είχαμε τέτοια παραδείγματα που σταματήσαμε τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων για ένα εξάμεινο και αυτό ήταν καταστροφή από πολλές άποψει. Και έδωσε πολύ άσχημο μήνυμα, ιδίω στη νέα γενεά. Άρα είμαστε και σε αυτό υπεύθυνοι. Επίσης υπεύθυνοι είμαστε για την ψηφιακή και ενεργειακή ένωση. Αυτό σημαίνει διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Υποδομές, τηλεπικοινωνίες, υποδομές τηλεπικοινωνιών. Η χρηματοδοτική προσπάθεια είναι διαρκής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρόγραμμα για τις βιομηχανικές περιοχές, για την ε, εκ νέου εκβιομηχάνηση περιοχών. Πολύ σημαντικά αυτά. Και θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα για του χρόνου και ειδική χρηματοδότηση. Αν και δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ακόμη. Τι, τι μορφή θα λάβει. Από τη δική μας σκοπιά πάντως θα είναι πολύ σημαντικό ομοίως. έξι το υπαθμό έξι λοιπόν ε, σχολείο μου. Αναφερθήκατε σε ορισμένους οργανισμούς όπως τον ASO και τη δυνατότητα χρηματοδότησης Πολύ σημαντικό αυτό για μας στη βάση των προσπαθειών που κάνουμε για να προχωρήσει η δέση μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Εκεί είμαστε υπεύθυνοι για 8-9 οργανισμούς στην Ένωση. Επαναδιάθεση ε, κονδυλίων από ένα τομέα σε άλλον. Να μην αποβεί σε βάρος υφιστάμενων έργων. Επίσης πολύ σημαντικό διότι το συζητήσαμε κάτι είπατε και εσείς σχετικά και χρειάζεται υποστήριξη τα προγράμματα αυτά, τα έργα αυτά. Τέλος, η Επιτροπή Ήτρε συμφωνεί με τις προτεραιότητές σας για τον προϋπολογισμό του 2018 και αναμένουμε βεβαίως πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν μας μένει πολύς χρόνος, όμως γνωρίζοντας τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή τα δημοσιονομικά όρια αν θέλετε επιθυμούμε ε, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν μια διαρκή χρηματοδότηση. Βεβαίως κοινωνική ασφάλεια σημαίνει δουλειές. Βιομηχανία, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις λοιπόν αυτές εκ μέρους μου που έχουν προκύψει και από συζητήσεις με τους συναδέλφους μου εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Αγαπητές και αγαπητοί, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν, λάβετε τον λόγο εφόσον το επιθυμείτε για να συμβάλλετε στη συζήτηση. Ε, Ο κύριος Τσέζακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρέμβασή σας και τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε, γιατί έτσι έχουμε μια ιδέα για τα προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για το 2018. Όπως ξέρετε, ε, τέλος Φεβρουαρίου οι Υπουργοί Οικονομικών ε, υιοθέτησαν συστάσεις για τον Ευρωπαϊκό Προβλογισμό και το 2018 και είπαν ότι θα επικεντρωθούν όπως και το 2017 σε αποτελεσματικές, αποτελεσματική ανταπόκριση στην ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη στήριξη των οικονομιών των κρατών μελών. Ο εισηγητής μίλησε για αυτά τα θέματα και ο Πρόεδρος επίσης. Και χαίρομαι που δεδομένων και των οικονομικών ε, ε, περιορισμών συγγνώμη, σε κάποια κράτη-μέλη, οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και οι πληρωμές θεωρητικά δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα βασιστούν στις πραγματικές ανάγκες. Όλα τα μέλη της ΣΥΤΡΕ ε, είμαι πεπισμένος ότι θα συμφωνήσουν ότι ως ε, τμήμα του προπολογισμού για το 2018 θα πρέπει να παράσχουμε χρηματοδότηση σε αυτό το επίπεδο ώστε αποτελεσματικά να υποστηρίξουμε την καινοτομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς επίσης και την ε, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει και την οικονομία την δημιουργία θέσεων, νέων θέσεων εργασίας, αλλά και άλλους στόχους που πρέπει να επιτύχει ο προπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Η συνέχιση των ε, τρεχόντων ε, ορίων, η άξιση τους παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ένωσης, είναι πραγματικά ε, ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία θα είναι σε τροχιά αναπτυξιακή και αυτό θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε με βιώσιμο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό δεδομένου και του σκελετού του προϋπολογισμού που έχουμε ήδη. Οπότε και η δική μας επιτροπή αλλά και άλλες επιτροπές νομίζω ότι θα δουλέψουν εντατικά για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί των στόχων του Κοινοβουλίου, αλλά και με το Συμβούλιο και βεβαίως εύχομαι στον εισηγητή κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Αυτό που λέτε ουσιαστικά αποτελεί συστάσεις σε μένα. Όταν θα ε, ε, συντάξω λοιπόν την επιστολή θα τη λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόταση αυτή να κάνουμε ανοιχτό διάλογο. Ε, χαιρετίζω την έμφαση που δίνετε κύριε συνάδελφε στην ανάπτυξη τους νέους και τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και την καινοτομία και την ανάπτυξη όπως είπες και εσύ Πρόεδρε. Ε, πρέπει όντως να μπορούμε να επενδύσουμε σε όλα τα στοιχεία της αλυσίδας κατανάλωσης και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη στο μέλλον. Τώρα για το Acer, θα απαντήσετε βεβαίως, αλλά το Acer προς το παρόν έχει αυξημένες αρμοδιότητες, χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται πόρους, για να μπορέσει να επιτύχει ακριβώς τους στόχους του και τις, να αρθεί στο ύψος των αρμοδιοτήτων του. Ε, καλωσορίζω την έμφαση που δίνεται στην ε, ε έμφαση στις επενδύσεις και στα πλαίσια του προγράμματος ε, ορίζοντας 2020, του ΣΕΦ και του ε, ε, και των υπολείπων προγραμμάτων. Ε, Βεβαίω, σε περίπτωση που η δική μου χώρα πιέσει για σκληρό Brexit, δυστυχώ δεν θα είμαστε μέρο τη ε, μακρόχρονη έρευνα που γίνεται ε, και που αποτελεί σημαντικής, ε, σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη τη της βιομηχανίας, της ιατρικής, για την έρευνα για την υγεία, την αντιμετώπιση ασθενειών όπω ο Καρκίνο, οπότε καλωσορίζω τι προτάσει σα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις και από μένα. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τις επενδύσεις και το, τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, έχουμε πολλούς ε, διαδρόμους, πολλά στοιχεία, πολλές ε, συνδέσεις μεταξύ του, βορού, βορρά και του νότου μέσω των αγωγών αερίου και μέσω της α, ε, τσιχικής δημοκρατίας αλλά και μέσω της Σλοβακίας και της Πολωνίας. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτά τα δύο στοιχεία δεν θα χαθούν στον προπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Δεύτερον, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στον προπολογισμό ε, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα υψηλής τάσης, γιατί είναι ουσιώδος σημασίας. Γνωρίζουμε ότι στην ε, Γερμανία ε, λείπουν οι υποδομές, οι σχετικές, δεν θέλω να, το, να επεκταθώ, είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά, οπότε θα πρέπει να δούμε τις διασυνδέσεις και μεταξύ άλλων χωρών κυρίως προς τα Βαλκάνια. Και τρίτον, μιλούμε για τις τεχνικές ε, εξελίξεις, γιατί και οι αεροπορικές μεταφορές αλλά και η πολιτική για το διάστημα είναι σημαντικά στοιχεία. Τα συζητήσαμε και πιο πριν για το πώς ε, θα ε, δομηθεί ε, ο ευρωπαϊκός διαστημικός χώρος στο μέλλον, αλλά και η ε, βιομηχανία ε, αεροπορικών μεταφορών επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη. Χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν, οπότε είναι σημαντικό να, υπάρξουν, να υπάρξει υποστήριξη από τον προπολογισμό για αυτούς τους τομείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δελίτσικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι για τα προκαταρτικά σχόλια του εισηγητού. Γενικώ νομίζω ότι έχει δώσει έμφαση στα σωστά στοιχεία. Είναι όντως ε, σωστές οι προτεραιότητες που έχει θέσει. Και νομίζω ότι καλύπτει και τις ανησυχίες της Επιτροπής μας. Συμπληρώνοντα τα σχόλιά σας, να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Και σε σχέση με τα άλλα χρηματοπιστωτικά ε, ε δημοσιονομικά εργαλεία. Μιλήστε για το ΕΦΣΙ και την ε, εκτίμηση που έχουμε όλοι. Ξέρουμε εις βάρος ποιων προγραμμάτων έχει δημιουργηθεί το ΕΦΣΙ Συμβαίνει βέβαια αυτό, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές πάντα, η επιτροπή μας δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ωστόσο, ας δούμε τον προπολογισμό αυτό για το κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, όχι το κατά πόσο είναι επιτυχή η ΣΟΕΦΣΗ, γιατί είναι, αλλά πόσο είναι επιτυχή σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Η δική μου η αξιολόγηση είναι αρκετά επικριτική. Για κάποιου τομεί, μάλιστα, θα έλεγα ότι η καινοτόμο φύση των ε, προγραμμάτων, ε, των project που έχουν χρηματοδοτηθεί, ε, είναι λίγο αμφισβητήσιμη. Τέλο πάντων, είναι συζητήσιμη. Δεν μπορώ να φανταστώ στο μέλλον οποιασδήποτε εξελίξεις να συμβαίνουν εις βάρος του ορίζοντα 2020 ας πούμε ή άλλου project και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά εντάξει αυτό είναι διαφορετικό θέμα γιατί κύριε Σιγητά δεν θα καταλήξουμε σε αυτό που είπατε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνιστική οικονομία χρειαζόμαστε ανάπτυξη, θέσεις εργασίας αλλά ο τρόπο αυτό δεν είναι ο σωστό για, να τα για να τα επιτύχουμε, ούτε μεσοπρόθεσμα ούτε πρόθεσμα. Οπότε, ούτε μακροπρόθεσμα. Οπότε αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Και επίση, σε σχέση με αυτό που είπατε για την δυνατότητα χρηματοδότηση των project από το 19% στο 13% μειώθηκε, ε, νομίζω ότι αυτό είναι προφανέ. Έχετε καλές προθέσεις νομίζω και όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις στις οποίες ε, αναφερθήκατε κι εσείς. Μιλήσατε για την ασφάλεια των πολιτών. Ο προπολογισμό δεν τον θυμάμαι βέβαια απ' έξω, αλλά νομίζω ένα 3% είναι αφοσιωμένο σε αυτό. Και ξέρουμε ότι ε, ίσως αυξηθεί. Δεν θα είναι λοιπόν εύκολο για εσάς στην όλη διαδικασία να εξασφαλίσετε ότι αυτή τη φορά δεν θα πληγεί η ασφάλεια των ε, πολιτών που είναι σημαντική για να προωθηθούν άλλες προτεραιότητες. Εμείς ήδη ήμασταν απογοητευμένοι από το πώς έγινε αυτό την προηγούμενη φορά, ελπίζω να μην ξαναγίνει. Τώρα για τα πιλωτικά προγράμματα, νομίζω ότι το, το μήνυμα είναι σαφές. Χαίρομαι που είναι και η Κομισιόν παρούσα, γιατί θέλω να κάνω ένα μονόπλευρο σχόλιο. Θα ήθελα η Κομισιόν να είναι πιστική σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που κάνει, γιατί εμείς το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. Θα μπορούσε κανείς να αμφιβάλλει για τις εκτιμήσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να είναι αμερόληπτη. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι έχει και αυτή τις δικές της προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και για το Acer, γιατί μας είπατε να κάνουμε τα σχόλιά μας, ε, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση σας. Το είπε και η Τερέζα, το είπε και ο Πρόεδρος. Δεν θέλουμε να υπάρξει ε, αύξηση της αλληλεξάρτησης εκεί, αλλά ο φόρτος εργασίας αυξάνεται στον Acer. Οπότε θα πρέπει να δούμε τους στόχους που έχει θέσει, οπότε εκ μέρους της Επιτροπής μας μπορώ να πω ότι θα το υποστηρίξουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο, ξέρω ότι ξεπερνάει λίγο αυτά που συζητούμε, αλλά Επειδή το σκεφτήκατε κι εσείς, θα ήθελα κι εγώ να το σχολιάσω. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Συμβούλιο. Κατανοώ ότι είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ ευαίσθητη με το Brexit, καταλαβαίνω ότι πρόκειται επίκυνται εκλογές, αλλά ε, εκλογές γίνονται σε όλα τα κρατημέλη μέσα στους επόμενους τρει-τέσσερι μήνες. Οπότε συμφωνώ ότι Υπάρχει απειλή των αρνητικών επιπτώσεων, αλλά θα πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να προχωρούμε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Τι θα κάνουμε, θα ζυγίσουμε το κάθε κράτος μέλος να δούμε ποιο είναι σε πιο δύσκολη εσωτερική θέση και ποιες ε, εκλογές σε ποιο κράτος μέλος είναι λιγότερο ευαίσθητες. Δεν θα το είχα θίξει γιατί ξέρω ότι είναι ευαίσθητο, αλλά δεν θα το είχα θίξει αν δεν το είχατε κάνει κι εσείς. Αλλά επειδή το είπατε ήθελα κι εγώ να προσθέσω κάτι. Αυτά λοιπόν πρόεδρε, συμφωνώ και με τα δικά σας σχόλια. Αναφερθήκατε κι εσείς σε κάποιες προτεραιότητε που δεν είναι στην αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Εμεί τονίζουμε τις δικέ μας προτεραιότητε, βέβαια, πλήρη στήριξη προς τον εισηγητή από μένα, αλλά θα περιμένουμε να κάνετε την θεωρία πράξη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά όλα τα σχόλια και για τον εισηγητή μας από την Επιτροπή Προπολογισμού αλλά και για μένα όταν θα συντάξω την επιστολή. Να ξαναδώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις καταρχάς. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν και από εσά, Πρόεδρε, και από τους συναδέλφους με την έννοια ότι η οικονομία δεν θα ενισχυθεί από μόνη της, ούτε θα λύσει τα προβλήματά της μόνη της. Οπότε οι βασικές προτεραιότητες πολιτικές που είχαμε τα τελευταία χρόνια και ήταν σωστά, σωστές ακριβώς λόγω και της αναδυόμενης φύσης που είχε η κατάσταση αυτή, ε, ε, ε, προσπαθήσαμε να διαθέσουμε όλες τους ε, Όλου του πόρου ε, για το Ταμείο της, για την Τουρκία για τους πρόσφυγε, για την Αφρική κτλ. Δεν μπορούμε πάνω λοιπόν να περιμένουμε η οικονομία να διορθωθεί από μόνη της, γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα της θέσης εργασία, την έρευνα, την κοινοτομία τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την νεολαία και τις σχετικές πρωτοβουλίες και, τα και το πρόγραμμα Εράσμους. Και όπως είπατε και εσείς, τα υπάρχοντα προγράμματα δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν. Συμφωνώ ότι το, προ... το το, δημοσιονομικό πλαίσιο το προωθήσαμε με βάση τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει. Τώρα, αν υπάρξουν νέες προτεραιότητες για την ασφάλεια ή για το, για το προσφυγικό, θα πρέπει να προσαρμόσουμε και εμείς τη θέση μας απέναντι στο Συμβούλιο, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, αλλά ίσως να χρειαστούν και φρέσκα κονδύλια γιατί αλλιώς θα επηρεαστούν τα υπάρχοντα project και συμφωνώ με τους, με τους συναδέλφους που λένε ότι η επαναδιάθεση δεν ε, ε, είναι σωστή προσέγγιση και για, γιατί τα υπάρχοντα προγράμματα δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν. Για το Brexit, το είπατε κι εσείς ε, σύντομα και εγώ είμαι εισηγητής για τον, εισηγητή, για τον προϋπολογισμό 2018. Το Brexit δεν πρόκειται να γίνει το 2018. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πλήρε μέλος της Ένωσης και το 2018, οπότε πλήρη δικαιώματα και πλήρε υποχρεώσει και στον τομέα της έρευνα. Τώρα το τι θα γίνει μετά ε, είναι ανοιχτό ακόμα. Έχουμε ε, ωφεληθεί από τη χρηματοδότηση ε, για την έρευνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πανεπιστήμια του επίση είναι πρώτη κατηγορία με εξαιρετικά ερευνητικά ιδρύματα. Οπότε αυτό που θέλουμε να δούμε για τον Brexit, μια που δεν θα γίνει του χρόνου, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει και καμία επίπτωση στον προπολογισμό. Τώρα, το τι θα γίνει μετά, θα το δούμε. Θα χάσουμε όντω ε, έναν συμβάλλοντα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και μετά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με τον προπολογισμό. Εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Στην Επιτροπή μα ήδη έχουμε αρχίσει να το μελετούμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν, υπάρχουν τρέχουσε συζητήσει για του ίδιου πόρου τη ε, Ένωση. με την προπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω βάρο για του ε, πολίτε, αλλά και ότι θα διατηρηθεί η σταθερότητα του ε, προπολογισμού μακροπρόθεσμα. Και για το ΕΦΣΥ, όπω είπα και στην αρχή, οι δύο εισηγητέ λένε να μην υπάρξουν ε, περαιτέρω περικοπέ. Αυτή είναι και η δική μου θέση. Ο κύριος, κύριε Τέλιτσκα, επειδή το ΕΦΣΙ δημιουργήθηκε με λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, είναι προ όφελό μα να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι επιτυχέ. Αν τώρα θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, χρηματοδότηση καινοτόμων project ή την αρεσιμότητα, τότε ναι, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν σωστό να υπά... Ναι, ω εργαλείο να κλείσει το κενό των επενδύσεων, αλλά βεβαίω θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσει αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητε. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτή είναι η αρχή του διαλόγου. Χαίρομαι που μπόρεσα να είμαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις και τα σχόλια που κάνατε. Όπως είπα η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους ε, σε όλη τη διαδικασία του, καθορισμού του προπολογισμού. Αυτά πρόεδρε από μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι που ήσουν μαζί μας σχεδόν για μία ώρα. Έχουμε και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Και φαντάζομαι ότι όλα όσα είπαμε θα ληφθούν και από αυτούς υπόψη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που θα υποβάλει σε μερικές εβδομάδες την πρότασή της. Οπότε θα θέλαμε, όσα αναφέρθηκαν σήμερα εδώ, να ληφθούν υπόψη και να φαίνεται αυτό και στην πρότασή σας. για την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Deadline for amendments on budget. προθεσμία για τις τροπολογίες για τον προπολογισμό 30 Ιουνίου 2017. Πιλωτικά προγράμματα 27 Απριλίου, ψηφοφορία της ΣΥΤΡΕ για τις γραμμές του προπολογισμού 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 18 και 19 και τα δύο μαζί. Εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, ηλεκτρικής ενέργειας, αναδιατύπωση του κανονισμού και κοινή κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οδηγία. Ένας κανονισμός και μία οδηγία. Θα τα δούμε από κοινού, όπως συζητήσαμε και αποφασίσαμε στη συνάντηση των συντονιστών πριν από κάποιους μήνες, και ο η και για τις δύο αυτές προτάσεις είναι ο Κρισιάνης Κάρινς. Να πω ο προτινόμενος, ότι ο προτινόμενος κανονισμός ε, ε, μιλά για, τα, για τη χοντρική πώληση και η ε, οδηγία για τη λιανική πώληση, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν στου ε, καταναλωτέ. Γι' αυτό θα τα δούμε από κοινού. Οι δύο προτάσει ε, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ του και γι' αυτό οι συντονιστέ τη ΣΥΤΕ, όπω είπα, αποφάσισαν να τι δούμε από κοινού. Οι ε, σκιώδει είναι οι ίδιοι και για, τα δύο, για τις δύο εκθέσεις. Ο στόχο είναι να εξχρονιστεί η ευρωπαϊκή αγορά, έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και να, να μπορέσει να επιτύχει και τους στόχους για το κλίμα, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη χρήση του ICT των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να είναι πιο αποκεντρωμένα και πιο αποτελεσματικά. Και βεβαίω υπάρχει και άμεση σύνδεση με την Ψηφιακή Ένωση, την ε, ε, Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Εκεί χρειάζεται σαφής ε, σημαντική χρηματοδότηση και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα νοικοκυριά θα μπορούν να έχουν φτηνή ηλεκτρική ενέργεια παντού στην Ευρώπη. Αυτές οι δύο προτάσεις, όπως είπα, συνδέονται άρρηκτα με άλλες 7 ε, προτάσεις του πακέτου για την ενέργεια και τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχουμε επιτάπητος κάποιες προτάσεις όχι καινούργιες, αλλά εν πάση περιπτώσει μια νέα προσέγγιση για, την, για το σχεδιασμό της αγοράς αερίου. Τώρα όμως θα μιλήσουμε μόνο για, το, για την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί βεβαίως Βέβαια όχι αποκλειστικά γιατί αν μιλήσουμε για την διαχείριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα μπούμε αναγκαστικά και στα νερά της αγοράς αερίου. Αυτά από μένα. Οπότε να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κρισιάνης Κάριν να α, παρέμβει. Οπότε θα του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να μιλήσει, γιατί θα μιλήσει για δύο σημεία. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα γενικό σχόλιο. Όλοι γνωρίζουμε πως ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά στον τομέα του ηλεκτρισμού, οπότε το παλιό μοντέλο μεγάλη παραγωγή, όπου όλοι είναι παθητικοί καταναλωτές ενώ, του ρεύματος ε, που προέρχεται από την κεντρική σταθμό, ε, που λειτουργεί είτε με φυσικό αέριο, είτε με πυρηνική ενέργεια, είτε με άνθρακα, έχει τελειώσει. Ανεξάρτητα αν τον θέλουμε ή όχι, η αγορά θα καθορίσει πια τα ε, ανανεώσιμες όλο και περισσότερο περισσότερο ώστε αυτές να αποτελούν πια τη βάση ενώ τα ορυκτά καύσιμα θα χρησιμοποιούνται όταν δεν έχει ε, αέρα ή όταν έχει πολύ συννεφιά ώστε να μην μπορούν ε, να λειτουργήσουν τα, ηλεκτρο... τα εργοστάσια. Ωστόσο ζούμε στον κόσμο των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν τις αγορές. με ολόκληρη τη δέσμη, αλλά ειδικά με αυτά τα δύο ε, ντοσιέ, θέλουμε να ε, μειωθούν οι τιμές ε, για τον τελικό καταναλωτή και θέλουμε να στείλουμε μηνύματα στους φορείς της αγοράς ώστε να κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις για να μπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής στην αγορά όταν αυτό χρειάζεται. Στις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, πρώτη φορά ασχολούμαστε πραγματικά με το κόστος, δηλαδή μείωση των τιμών μέσω αυξημένου ανταγωνισμού και μέσω ορθής λειτουργίας των αγορών. Θέλω να αναφερθώ σε τέσσερα κυρίω ζητήματα, όπου πιστεύω ότι αυτοί οι δύο φάκελοι θα παίξουν βασικό ρόλο. Το ένα είναι οι δυνατότητες παραγωγής που διασταυρώνονται με τις επιδοτήσεις. Το δεύτερο είναι οι συνεργασίες το τρίτο είναι οι περιοχές ε, ε, διαγωνισμών και μετά έχουμε την λειτουργία της αγοράς με τις δυνατότητες ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή το, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τι είδους ε, αποθεματικό χρειάζονται. Αυτό το αποφασίζει το κάθε κράτος. Η Κομισιόν προτείνει να υπάρχει πρώτα μία περιφερειακή αξιολόγηση ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες ε, για έναν τέτοιο μηχανισμό. Η Κομισιόν θέλει δηλαδή να ξεπεράσουμε τα σύνορα των κρατών μελών για να ορίσουμε αν θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Τι, είναι τώρα αυτοί οι μηχανισμοί αποθήκευσης. Κατά κάποιο τρόπο είναι ε, επιδοτήσεις που εμείς ως καταναλωτές πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Είτε ο καταναλωτής είναι η βιομηχανία, είτε είναι ένα ε, σπίτι, ένα νοικοκυριό. Εμείς θέλουμε αυτοί οι μηχανισμοί να ε, διατηρούνται σε ένα μήνυμα και να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική. Όταν, ας πούμε, η αγορά δεν έχει αρκετό ηλεκτρισμό. Πρέπει να υπάρχει και μια διασυνοριακή διάσταση σε αυτούς τους μηχανισμούς αποθήκευσης, γιατί έτσι όπως αναπτύσσεται η αγορά, ο ηλεκτρισμός ήδη περνά τα σύνορα, δεν είναι κάτι που ανήκει στο απότερο μέλλον. Αν βλέπουμε λοιπόν τους μηχανισμούς αποθήκευσης, ένα είδος αποθεματικού ώστε διαρκώς να έχουμε αναμένα τα φώτα μας, Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την περιφερειακή διάσταση. Η Κομισιόν προτείνει επιλεξιμότητα για τους μηχανισμούς αποθήκευσης που συνδέονται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, φαντάζομαι ότι θα έχετε να πείτε πολλά γι' αυτό, αλλά πάντως πρέπει να το δούμε από την πλευρά της ασφάλειας ανεφοδιασμού, της σκοπιμότητας και της επικορικότητας. Το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Το δεύτερο θέμα είναι η περιφερειακή συνεργασία στα περιφερειακά κέντρα στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους RSCs που είναι οι περιφερειακοί συντονιστές. Τώρα αρχίζουν να λειτουργούν στο κράτος μέλος μου και στα Βαλκάνια. Αυτό θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιανουάριο όπου θα λειτουργούν ε, συνδεδεμένοι. Δηλαδή είναι ένα είδος συντονισμού ανάμεσα στα συστήματα να είμαστε μάλλον στους ε, φορείς ε, διαχείρισης ε, των συστημάτων διαβίβασης ή μεταφοράς. η Κομισιόν προτείνει αυτά τα, αυτοί οι περιφερειακοί συντονιστέ να αντικαταστήσουν του εθνικού ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καλύτερου υπολογισμού για την ε, δυνατότητα τη αποθήκευσης, τις ανάγκες κτλ. Δικό μου σχόλιο ότι ναι, για να μπορεί να λειτουργήσει η αγορά πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα και σε περιφερειακό επίπεδο. Όμως ρωτώ με. Όμως οι αρμοδιότητες πώς θα μοιραστούν. Αυτή τη στιγμή οι κρατικοί ρυθμιστές είναι αυτοί που φέρνουν όλη την ευθύνη που σε κάποιες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε ένα κράτος μέλος, ενώ σε κάποιο κράτος μέλος υπάρχουν και περισσότεροι από έναν TSO, δηλαδή τοπικοί συντονιστές. Πρέπει ωστόσο να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Τρίτο, ε, οι περιφέρειες ε, για τις ε, προμήθειες. οι τιμέ που ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τη συμφόρηση. Υπάρχουν κράτη-μέλη δηλαδή, και σκέφτομαι ένα συγκεκριμένα, όπου υπάρχει εσωτερική συμφόρηση, ενώ υπάρχει μόνο μία τιμή, αντί να αφήσουμε ε, την συμφόρηση να δείξει ποια είναι η προσφορά και ποια η ζήτηση. Η Κομισιόν προτείνει οι ζώνες αυτές να ορίζονται από διαρθρωτικές ε, ζώνες που θα περιορίζονται ε, από τις περιοχές όπου δεν υπάρχει συμφόρηση, δηλαδή μέχρι τα σύνορα σε μια ιδανική αγορά αυτό θα ήταν ε, απλό. Δεν ήταν όλα πολύ καλά συνδεδεμένα, δεν θα υπήρχε πουθενά σημείο συμφόρηση και όλα θα λειτουργούσαν ομαλά. Αυτά είναι όνειρα θερινή νυχτό. Είναι μια ιδανική κατάσταση. Όμω αυτό που έχουμε εμεί να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι ε, μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Η ζώνες τιμών είναι σημαντικές για να έχουμε τι απαραίτητε επενδύσεις. Αν ας πούμε η τιμή σε κάποιο σημείο της Ευρώπης, ε, η τιμή θα πρέπει να είναι ψηλή εφόσον υπάρχει χαμηλή προσφορά και μεγάλη ζήτηση. Αλλά αν αυτό το κομμάτι της Ευρώπης βρίσκεται σε μια ζώνη τιμών που δείχνει ότι τεχνητά η τιμή είναι πιο χαμηλή από ό,τι θα έπρεπε, τότε δεν θα γίνονται επενδύσεις, δεν θα υπάρχει κίνητρο για κανέναν να φτιάξει ε, διασυνδέσεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα για τις επενδύσεις. Και τέταρτον, η ζήτηση η ζήτηση από πλευράς των καταναλωτών ε, σε σχέση με τις ε, τιμές και την παραγωγή ενέργειας. Αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος παράγει την ενέργεια και σήμερα πολλοί καταναλωτές ε, στα νοικοκυριά έχουν ακόμα Ωστόσο, ρυθμιζόμενες τιμές. Αν θέλουμε να γίνει ενεργειακή μετάβαση, να περάσουμε από τα, από τα ορυκτά καύσιμα σε λιγότερο ρηπαίνουσε πηγέ, όπως η βιομάζα και σε κάποιο βαθμό ύδρο ε, είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Οπότε θα φυσήξει ο αέρας, θα λάμψει ο ήλιος, αρκετά. Έχουμε κειμενόμενη, κειμενόμενη ε, προσφορά. Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να παράγουμε ενέργεια όταν το παραπάνω τον, χρειαζόμαστε, ενώ οι καταναλωτές να μπορούν να μειώνουν τη χρήση όταν υπάρχει πολλή ζήτηση. Και έτσι πρέπει να έχουμε και τεχνολογία σε επίπεδο νοικοκυριού. Εάν δηλαδή μπορέσουμε να εμπλέξουμε τον καταναλωτή, μπορεί να χρειαζόμαστε λιγότερο την αποθήκευση ε, ηλεκτρισμού στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ζουμί. Ευχαριστώ. Βέλνερ τώρα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πακέτο για την καθαρή ενέργεια περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς φακέλους. Κατά την άποψή μου, ο κανονισμός και η οδηγία θα πρέπει να να τους δοθεί μια πολύ σημαντική έμφαση γιατί εδώ μιλούμε για, το νέο, για τη νέα δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει αλλάξει αυτή τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός των εμπλεκόμενων φορέων στην αγορά έχει αυξηθεί είτε ως παθητικοί καταναλωτές έχουν αυξηθεί επίσης, αλλά και η αποκέντρωση των, της παροχής επίσης έχει ε, διαφοροποιηθεί και η δομή τη μελλοντική αγορά ηλεκτρικής ενέργεια θα πρέπει αυτά να τα λάβει υπόψη στο μέλλον. Τώρα για την επιμέρους σημεία υποχρεώσει υποχρεώσεις των διαφόρων φορέων στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια, του προμηθευτέ, του διανομή, τι εθνικέ νομιστικές αρχέ, αλλά κυρίω του καταναλωτέ θα πρέπει να του λάβουμε υπόψη και θα πρέπει όλε αυτέ τι εξελίξει των τελευταίων ετών, να τι εντάξουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτέ. Οι σημαντικοί παίκτες στις αγορές του μέλλοντος θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ε, δυνατότητα επιλογής και σε παροχή ενέργειας και σε δυνατότητα εξορρόψης ε, τιμών και σε καλλιέργεια, ε, παραγωγή ενέργειας αλλά και πώληση αυτής. Άλλο ένα σημαντικό σημείο για το νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να, έχει, να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια στο σύστημα αλλά και ασφάλεια στην προμήθεια. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη διασυνοριακή συνεργασία, πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα ώστε να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια στην προμήθεια και να είναι αυτή και φτηνή όσο δυνατόν γίνεται και για την βιομηχανία και για τον καταναλωτή. Πέραν αυτού, ως κοιότηση συγγήτρια, θα ακολουθήσω μια ε, προσέγγιση αγοράς ε, αμυγός ενεργειακής. Προς το παρόν υπάρχουν ε, περίπου 13 κρατημέλη που έχουν διάφορους μηχανισμούς και οι τρέχοντες, υπάρχοντες μηχανισμοί κατακαιρματίζουν την αγορά αντί να την διασυνδέουν πιο πολύ. Και είμαι πεπισμένη ότι η πιο στενή διασυνοριακή συνεργασία θα βοηθήσει στην καλύτερη παραγωγή ενέργειας, θα βοηθήσει τα δίκτυα διανομής και παραγωγής έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει αρκετό ρεύμα για όλους όπου και αν βρίσκονται και ότι δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα ή αδιέξοδα. Αυτοί οι μηχανισμοί δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι, αν υπάρχουν, μόνο διασυνοριακοί και θα πρέπει να είναι και η τελευταία λύση. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και με έχει απασχολήσει πολύ είναι το θέμα των ζωνών, των τιμολογικών ζωνών. Ε, η Κομισιόν κάνει μια πρόταση για τα δίκτυα μεταφοράς. Η, η πρόταση της Κομισιόν όμως έχει ως αποτέλεσμα η Γερμανία ας να χωρίζεται σε δύο ζώνες. Και αυτό δεν είναι δυνατό να συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την, ε, να αποφασίζει για τις ε, ζώνες τιμολόγησης οι οποίες είναι κατεξοχήν ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και με τους άλλους συναδέλφους αλλά και με τον εισηγητή για να έχουμε στο τέλος μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Βαϊσάκα που αντικαθιστά τον κύριο Κρασνοδέμσκι, εξ ονόματος του ΙΣΙΑΡ. Ο κύριος Τσέσακ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, αντικαθιστώ τον κύριο Κρασνοντεύσκη που είναι ο σκιώδης εισηγητής και θα σας ε, παρουσιάσω τη δική του γνώμη και κατά συνέπεια της ομάδας μας. Δεν μπορούσε να είναι, βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά ήθελε να υποβάλει τα αρχικά του σχόλια για αυτή την πρόταση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος στόχος της Ενεργειακής Ένωσης είναι η εγγύηση των σταθερών, ε, της σταθερής προσφοράς σε προσιτές τιμές. Αυτό αναφέρεται και στον ηλεκτρισμό. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ανεξαρτησία τους ε, ως προς αυτό το θέμα. Γι' αυτό και η ιδέα της περιφερειοποίησης της αγοράς είναι επικίνδυνη, γιατί είναι πιθανό ε, πολλές, Ε, να χαθούν, γιατί δεν συμμορφούνται προς τις υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Όσον αφορά την εισαγόμενη ενέργεια, μπορεί αυτό να βασίζεται, να, να σημαίνει μάλλον τους κύριους ε, ε, παραγωγούς, δηλαδή Γερμανία και Γαλλία. Εάν χρειαστεί κάποιοι χρήστες να, χρήστες να σβήσουν, Ε, ποιες θα είναι οι λύσεις για να προβλεφθεί και να καταπολεμηθεί η ενεργειακή ένδυα. Οι περιφερειακές λύσεις μπορεί να λειτουργήσουν αν οι χώρες δεν εξαρτώνται από κάποιον πολύ ισχυρότερο εταίρο. Να συνεχίσουν δηλαδή να έχουν τη δική τους παραγωγή οι χώρες, ακόμα και αν αυτή χρησιμοποιείται ε, μόνο σε περίπτωση μείωση τη προσφορά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας ε, συμπεριλαμβανομένη τη παροχή ηλεκτρισμού προς τους καταναλωτέ είναι υποχρέωση που βαραίνει τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν μακροπρόθεσμα την ανεξαρτησία τους και την δυνατότητα παραγωγή ηλεκτρισμού. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, ε, για τα σχολιά σας και η κυρία Νινάρ που αντικαθιστά την κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Καΐα Κάλλας, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα. Καλωσορίζει αυτή την αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού, που είναι απαραίτητη αν θέλουμε να διηγηθούμε του αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών και να δώσουμε επίσης, να προσφέρουμε χαμηλότερες τιμές στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή η αγορά ε, βασίζεται σε κεντρική παραγωγή ε, δεν, ε, δεν προσαρμόζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ούτε ανταποκρίνεται στο επίπεδο ευελιξίας που χρειάζεται σήμερα. Πιστεύει επίσης ότι στην εργασία μας για την αναθεώρηση αυτών των προτάσεων, καλό είναι να βασιστούμε στις ήδη υπάρχουσες ε, καλές πρακτικές, όπως για παράδειγμα το North Pool Market. Εάν δεν θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μια αυξανόμενη διαφορά ανάμεσα στην Νότια Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να διατηρήσουμε αυτό τον στόχο υπόψη μας, ώστε να κατά την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης για τις ε, αγορές ε, ε, ε θα πρέπει αυτοί, αυτοί οι μηχανισμοί παραγωγής να μην στρεβλώνουν την αγορά ε, και να δούμε κατά πόσο αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αρκούν, γιατί εφόσον δημιουργούνται αυτές οι αγορές είναι πολύ δύσκολο κανείς να μην τις χρησιμοποιήσει, από ότι να μην τις φτιάξει καν για την ελληνική πώληση, εάν η χονδρική πώληση καταστεί πιο ευέλικτη, είναι σημαντικό η ευελιξία να περάσει και στη ελληνική αγορά, ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές. Γι' αυτό το να δημιουργηθούν κίνητρα για τη ε, τιμολόγηση είναι καλή λύση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και ένα phase-out για τις ρυθμιζόμενες τιμές, γιατί αυτό προκαλεί στρεβλώσεις εις βάρος του καταναλωτή. Ωστόσο, η βελεξία δεν μπορεί να είναι η μέγιστη στην ελληνική αγορά, αν οι καταναλωτές δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, την απαραίτητη ενημέρωση. Και δεν μιλάμε για μια το χρόνο ή μια φορά τους έξι μήνες, αλλά να έχουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο που θα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται την καθημερινή του τους κατανάλωση. Η Κομισιόν ε, τονίζει ότι τα οι ευφυείς μετρητές έχουν προγραμματιστεί μόνο για 17 κράτη-μέλη, άρα δεν αρκούν. Επιπλέον, οι λύσεις συζήτησης και προσφοράς θα αναπτυχθούν εάν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγορά και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για καινοτομία στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα τις καινοτομίε που βασίζονται στα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την κυρία Κάλλας να φτιάξουμε νέες νέες τεχνικές που μπορεί να συμβάλλουν σε πιο αποτελεσματικές αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ και η κυρία Κάλλας προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και τους συναδέλφους για αυτά τα δύο θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Και τώρα ο κύριος Τούρμες, εξ ονόμαστον των Πρασίμων. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Γέρση. Η αγορά μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη μου όταν έχουμε το πραγματικό κόστος. Και μια πτυχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι αν όλοι πληρώνουν για την ρήπανση, αν όλοι πληρώνουν για τα απορρίμματά τους και αν όλοι πληρώνουν για τον ε, κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Νέες δυνατότητες ε, πληρωμής είναι μια επιπλέον στρέβλωση και είμαι ευτυχής που εδώ βλέπω ότι έχουμε πλειοψηφία στο να λέμε ότι έχουμε άκαμπτη υπερπαραγωγή στην ε, Ευρώπη. Και θα μπορούσαμε ίσως και να ενισχύσουμε το κείμενο που έχει προτείνει η Κομισιόν. Δεύτερον, χρειάζεται να παράσουμε από την ακαμψία στην ε, ευληγησία, στην ευελιξία. Η σημερινή αγορά είναι άκαμπτη, ενώ αντίθετα χρειαζόμαστε ευελιξία, ευέλικτα εργοστάσια παραγωγής ε, και ούτω καθεξής. Και βέβαια κάθε ε, ατομικό πλυντήριο ρούχων μπορεί να παίξει ρόλο αν το δούμε σε βάθος 20 χρόνων, ενώ εγώ προτείνω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα κτίρια, τα γραφεία και μετά να κινηθούμε στο μικρότερο, χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε με τους μεγάλους καταναλωτές και να βάλουμε εκεί περισσότερη ευελιξία. Τώρα, περιφερειακές αγορές. Η μουσική παίζει όχι για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η γερμανική αγορά δεν υπάρχει πια. Η γαλλική αγορά επίσης και ευτυχώς γιατί αν υπήρχε φέτος το χειμώνα η Γαλλία θα έχει πέσει στο σκοτάδι, θα έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Αυτό που χρειάζεται είναι ε, σχηρές περιφερειακές αγορές, North Pool, κεντρική, ανατολική και πρέπει επιγόντως να φτιάξουμε μια περιφερειακή αγορά για την Νότια Ευρώπη που πράγμα που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Θετικέ επιπτώσει για του καταναλωτέ στη Νότια Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν αυτό να το αντικατοπτρίσουμε. ποιο ρυθμίζει τις περιφερειακές αγορές και Νομίζω πως δεν μπορείς, να, να μην έχεις έναν εθνικό διαιτητή όταν είναι περιφερειακή αγορά. Χρειάζεται περιφερειακή αγορά, αλλά χρειάζεται ο συγκεκριμένος ρόλο για το ΆΙΣΕΡ, για την Κομισιόν, να υπάρχει ένα καθρέφτη τη πραγματική αγορά. τιμολόγηση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα όπως στην Καλιφόρνια με μικροαγορές που με πολύ μικρή ρευστότητα ή μπορεί να έχεις κάποιες φορές πράγματα που δεν λειτουργούν ε, ομαλά και όλοι πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε ότι η Γερμανία έχει πρόβλημα. Αλλά η Γερμανία έχει αρχίσει να λύνει και το πρόβλημα με κάποια καθυστέρηση. Δεν θέλω να πάω στο Βαβαρία και γιατί και έχουν καθυστερήσει τα κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται μια μέση λύση. Πρέπει να πιεστούν χώρες όπως η Γερμανία να δώσουν τα δίχτυά τους. Και η τιμολόγηση έχει νόημα, αλλά όχι μικροτιμολόγηση. Χρειάζεται μεγάλες ρευστές αγορές, ώστε να έχουμε και μεγάλες ρευστές αγορές με, με προϊόντα 50, 30, 5 λεπτά. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσουν με χαμηλό κόστος καλύτερα οι αγορές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Yeah, Ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε. Με τον κανονισμό και την οδηγία έχουμε προτάσεις στο τραπέζι που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο σχεδιασμός της αγοράς ρεύματος αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένα σύστημα στέρεο, σταθερό και κυρίως που να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο γίνεται περισσότερο. Με πρώτη ματιά, στους δύο φακέλους μας απασχολεί το εξής. Πρώτο, η διαδικασία τροφοδότηση, Τη συζήτηση έχουμε ξανακάνει. Για μας στη Γερμανία ήταν σημαντικός παράγοντας ανάπτυξη για τι ανανεώσιμε ενέργειε. αυτό. Η δυνατότητα δηλαδή του ιδιότητα να τροφοδοτεί το ρεύμα που του περισσεύει στο δίκτυο. Να διατηρηθεί λοιπόν αυτό. Αυτή είναι η θέση μα και δεν είναι νέα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή, σωστά στοχευμένη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όριο 500 κιλοβατόρων. Κιλοβάτ μάλλον. Πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει λοιπόν να περιληφθεί η δυνατότητα τροφοδότησης και άνω των 500 κιλοβάτ. Να μην χαθεί αυτό το πλεονέκτημα. Αυτό ζητούμε εμείς. Επίσης, θεωρούμε ότι μέτρα με αναδρομική ισχύ και νομικά και επισουσίας είναι προβληματικά. Πρέπει να εξετάσουμε και τις άλλες προτάσεις στη μορφή θα λάβουν. Τι αποτέλεσμα θα έχουν. Δική μας ανησυχία είναι και είναι γνωστό αυτό, ότι ίσως έχουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πάντως, να διεξαχθεί συζήτηση. Γενικά, η πάυση λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας, εφόσον απαιτείται, μόνο εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση. Από την άλλη μεριά πρέπει να είναι σαφές επίσης ότι κλείνουν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας για να έχουν προτεραιότητα οι παραδοσιακέ Μεγάλο πρόβλημα αυτό για μας. Και αυτό γνωστό είναι. Στο άρθρο 12 νομίζουμε πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι διαχειριστές των δικτύων είναι υπεύθυνοι και για την επέκταση του δικτύου και για την συμπερίληψη περισσότερων πηγών ανανεώσιμης ε, ενέργειας. Το άλλο είναι για ε, τις ε, ικανότητες για τις χωρητικότητες της αγοράς Εμεί είδαμε ποια είναι η διατύπωση του εισηγητού διαμεθοριακά και ότι πρέπει να γίνεται περιφερειακή αξιολόγηση και άλλα τέτοια σχετικά. Ναι, να δούμε όμως πώς θα διαμορφωθούν οι λεπτομέρειες. Η αγορά ικανότητας δεν είναι ο σωστός δρόμος όπως το διατυπώνεται. Τώρα να οθούνται παραδοσιακές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε, ένα ανταγωνισμό, τότε αν θέλετε να γίνει αυτό θα πρέπει να πάψουν και οι επιδοτήσεις για τον άνθρακα και άλλες παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 23 να μπορούν να παράγουν μέχρι 550 ε, γραμμάρια, ε, ε, κυβικό μέτρο κλπ. ή τα νέα εργοστάσια καύση άνθρακα. Σύμφωνα πρέπει να υπάρχει, σύμφωνα, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και να γίνει προσπάθεια επίσης ο κανονισμός, εφόσον τεθεί άμεσα σε ισχύ, να ισχύει για όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Γίνονται προτάσεις και για τις Πράγματι θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Για τις τιμές θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αρκούμε σε αυτά. Much, Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο κύριος Ταμπουράνο της ομάδας EFDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων που αφορούν την αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Για διάφορου λόγου, αυτοί οι κανόνε που διέπουν τώρα την αγορά ηλεκτρισμού δεν ε, συνάδουν με τι δεσμεύσει που αναλάβαμε στο Παρίσι. Ελπίζω πω θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εργασία του εισηγητή ώστε να υπάρξει η περιφοριοποίηση, η ευελιξία, η διαφοροποίηση και ή πολιτικές, ή εθνικές από την άλλη πλευρά. Το σημείο κίνησης που μας προσφέρει η Κομισιόνα περιλαμβάνει διάφορα θετικά στοιχεία ε, που πάντως εμείς θα πρέπει να τα ενισχύσουμε. Η κεντρική θέση του καταναλωτή, η ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση για την εισαγωγή μηχανισμών αποθήκευσης δυνατοτήτων, η δυνατότητα ανάπτυξης των υπηρεσιών ενέργειας, η ε, διακύμαση των τιμών σε σχέση με τη ζήτηση. Θέλουμε το σύστημα να, είναι όσο, να, γίνει, να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα 100% ανανεώσιμο και γι' αυτό θα πρέπει ο εισηγητής κατά τη γνώμη μας να λάβει υπόψη τέσσερα ζητήματα που θεωρώ ε, προτεραιότητας. Να συνεχίσει η αγορά να λειτουργεί χωρίς αυτή τη μόνιμη υπερπαραγωγικότητα τα 550 γραμμάρια ε, διοξιδίου του άνθρακα ανά κιλοβατόρα θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλό κατόφλι σε σχέση με την παροχή επιδοτήσεων και ακόμα προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιο είναι το σημείο, καλύτερο σημείο κίνησης. Ο συνάδελφος της ΓΟΕ πρότεινε μια συγκεκριμένη τιμή. Πάντως, όποια και θα είναι τελικά αυτή η τιμή, θα πρέπει να μειούται ε, με την πάροδο του χρόνου. Η Κομισιόν επεξεργάστηκε ένα σύστημα εντοπισμού των πιο αποδοτικών τεχνολογιών στο πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές και νομίζω πως θα πρέπει σε αυτό να κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά έτσι ώστε ή ε, τα εργοστάσια ε, παραγωγής να σέβονται και τα στάνταρ ποιότητας του αέρα. Εάν θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στους στόχους του Παρισιού, θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα είναι ανοιχτοί σε κάθε πηγή που υπάρχει και θα είναι συνεπείς με την ε, Εξάλληψη της χρήσης του άνθρακα. Το να αποφύγουμε τώρα οποιοδήποτε είδος επιδότησης για τους παραγωγούς ενέργειας με το ε, επί ότι αυτοί ε, αποφασίζουν τον όγκο ενέργειας που θα παράγουν με βάση την κατανάλωση. Αν θέλουμε ο καταναλωτής όμως να ε, καταναλώνει καλύτερα και λιγότερο και το ΜΕΓΑΒΑΤ θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις τιμές. Άρα τι νόημα έχει να υπάρχουν ομαδοποίησεις να υπάρχουν ε, εταιρείε ενέργεια όταν μετά αφήνουμε ανοιχτό την πόρτα για επιδοτήσει ή αντισταθμίσει σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα ήθελα να τιμωρείται αυτό που προσφέρει καινοτόμε υπηρεσίε στην οπτική ανταπόκριση των ε, κλιματικών στόχων, να μην παραμείνει δηλαδή ανοιχτό το παραθυράκι για την υπερεκμετάλλευση του τομέα. Σημείο 4, 17, ε, άρθρο 17 αναφέρομαι. Τώρα, ανανεώσιμες. Εφόσον δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν... Ε, ε, μάλλον θα πρέπει να μπουν στο ίδιο επίπεδο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τις παραδοσιακές. Και επίσης υπάρχουν, υπάρχουν κίνητρα ώστε να προωθηθούν νέοι φορείς στην αγορά σε σχέση με τη μείωση της, ε, των απολειών ε, ε, διαβίβασης, μεγάλη και καλύτερη διαχείριση των δικτύων, περισσότερη ευελιξία και καλύτερη ευελιξία. Ιδιαίτερα τα, συστήματα, τα κλειστά συστήματα διανομής θα πρέπει να προωθηθούν για όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη για το δίκτυο το ενεργειακό εν γέννη. Επίσης, η ρήπη του φαινομένου του θερμοκηπίου να μείνουν κάτω από τα όρια του Παρισιού, δηλαδή να παραμείνει ένα ισότιμο πεδίο για όλους τους παίκτες της αγοράς, όπως λέει και η Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδησίδες. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Πρώτος ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Δύσκολη έκθεση αυτή και μπράβο σας. Η έκθεση την να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της που είναι οι φιλόδοξες αλλά δεν έχουν εξεγηθεί απαρκώς. Πιο συγκεκριμένα πώς θα βρεθεί ένα μοντέλο που θα λειτουργήσει σε 27-28 χώρες μέλη. Ελπίζω τώρα με την ευκαιρία της επόμε, των επόμενων επικειμένων εκλογών η Μεγάλη Βρετανία να αλλάξει άποψη για το Brexit. Αλλά ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα της Ρουμανίας. Για να μην λέμε και πολλά λόγια. Μηχανισμός αντιστάθμισης που δημιουργείται όταν δεν μπορούν να παράγονται ανανεώσιμες ενέργειες. Επειδή, για παράδειγμα, οι υποσυνθήκες χειμώνα μπορεί να σταματήσουν οι αιωλικές γεννήτρες ή μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη χιονόπτωση άρα δεν υπάρχει ούτε ηλιακή ενέργεια. Άρα μένουν μόνο τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος από άνθρακα, που είναι μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενέργειας. Ποιος θα παράγει την ενέργεια στη Ρουμανία εάν γίνει δεκτό το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Υπουργείο Ενέργειας στη Ρουμανία λέει ότι είναι αδύνατον. Όταν λέω ότι είναι αδύνατον, εννοώ ότι με τέτοιες χειμερινές θερμοκρασίες πάρα πολύ χαμηλές, το πρώτο δωδεκάωρο αυξάνεται κάθετα η θνησιμότητα ηλικιωμένων προσώπων. Να μην σας πω τι γίνεται στις 24 ώρες και παγώνουν ολόκληρα κτίρια και όλες οι εγκαταστάσεις τους. Αυτά τα πράγματα πάντα σκεφτούμε πολύ καλά και να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα ο μηχανισμός που προτείνεται, ώστε να μην παραμείνει ουτοπικός και να προσφερθεί ταυτόχρονα η ασφάλεια λειτουργίας Δεύτερο, να προσέξουμε ιδιαίτερα τα περιφερά κέντρα. Υπάρχουν σήμερα οι ευθύνε των χωρών μελών μέσα από τα εθνικά τους κέντρα. Αν τώρα μεταφερθούν οι ευθύνε σε επίπεδο που δεν διαθέτει ούτε την ε, ε, ε, τεχνική επάρκεια αλλά ούτε και το επίπεδο ευθύνη, θα προκαλέσουμε προβλήματα. Δεν πρέπει να προκαλέσουμε σύγχυση και στις εθνικές αγορές ενέργειας διότι πολλές χώρες μέλη πολλούν ενέργεια. Δεν μπορούμε να συγχέουμε τις αγορές με την διασφάλιση της παροχής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε μια τέτοια προσέγγιση, η οποία έχει πολλές θετικές πτυχές, πρέπει να προσέξουμε ορισμένες λεπτομέρειες όπως αυτές που προανέφερα, που μπορούν να καταστρέψουν την ίδια τη ουσία της εκθέσεως, διότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Ιδίω επειδή σήμερα δεν έχουμε τρόπους να αποθηκεύσουμε την παραγόμενη ενέργεια. Μια εγκατάσταση υδροελεκτρικής ενέργειας που κοστίζει εκατομμύρια ευρώ δεν διαθέτει όμως τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την παραγόμενη ενέργεια. Άρα χρειάζεται να βρούμε τεχνικές λύσεις. Με μια οπτική των επόμενων 20 ετών. ώστε να μπορέσει να υποστηριχτεί το περιεχόμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Λίγα σχόλια. Πρώτα γενικού χαρακτήρα συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Νίκα που τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Βεβαίως όλοι θέλουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας, όμως οι αγορές αναχώρα είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στον νέο αυτό σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και χρειάζονται και οι capacity markets, θα τις χρειαστούμε δηλαδή και μεσοπρόθεσμα. Μακάρι να μην τις χρειαζόμαστε, να τις χρειαζόμαστε όμως ακόμη για να διασφαλίσουμε αυτό που με απασχολεί εμένα για παράδειγμα είναι κυρίως η ασφάλεια της παροχής ενέργειας και αν τη θέσουμε σε κίνδυνο να μην μπορούν να τροφοδοτούνται δηλαδή με ενέργεια οι βιομηχανίες μας αυτό σημαίνει και τεράστια ζημιά για την οικονομία. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να εξεταστούν οι προτάσεις της Κομισιόν με τους μηχανισμούς παραγωγικής ικανότητας. Διότι μέσω και μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουμε να στερηθούμε τους μηχανισμούς αυτούς. Μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποιες βασικές αρχές, αλλά θεωρώ ότι από τώρα ήδη θα χρειαστούμε το status quo αυτό για να κινηθούμε και προς την κατεύθυνση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την ανάπτυξη των δικτύων και επέκταση των δικτύων σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερο σημείο για, τον, για τους μηχανισμούς ικανοτήτων, capacity mechanism. Δεν θα πρέπει να να φαινός ανάμεσα στα κριτήρια των εξοικονομήσεων του στόχου 1 και στην εντατικοποίηση από τη, μια, από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά την ασφάλεια της παροχής ενέργειας. Θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σταθμοί παραγωγής ενέργειας εργοστάσια τα οποία να μην ξεπερνούν τα 550 γραμμάρια ε, διοξιδίου του άνθρακος ανά κιλοβατόρα. Ε, το όριο αυτό δεν μπορεί να ισχύσει ακόμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπορεί να, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή εφεδρικής χρήσης τους των εργοστασίων αυτών. Έχουμε άλλα εργαλεία. Έχουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών, για παράδειγμα. Να μην συγχέονται οι πλευρές αυτές. Τέλος, το άρθρο 13 του κανονισμού. Νομίζω ότι πάντως η δική μου σκέψη είναι ότι η κατανομή των ζωνών πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη για να εξασφαλίζεται μια εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες της αγοράς για να μπορούν να λαμβάνονται και αποφάσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να μην διακυβεύονται αυτές. Είναι σημαντική λοιπόν, είναι σημαντικός σχεδιασμός των ζωνών κατανομής να γίνει με συμφωνία όλων και με επαρκή μεταβατική περίοδο. Σημειώνω δηλαδή ότι Χρειαζόμαστε την κατανομή ζωνών. Μακάρι να μην το χρειαζόμασταν, αλλά η πραγματικότητα είναι όπως είναι, η εξελίξη είναι όπως είναι. Και χρειάζεται και ένα σενάριο μεταβατικό και γι' αυτό νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν μπορεί να παραμείνει να ανατεθεί μάλλον η απόφαση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Γκρίφιν. Ευχαριστώ. Ο σχεδιασμό τη αγορά είναι πραγματικά ουσιώδη σημασία φάκελο που θα ορίσει το μέλλον τη μετάβαση ε, τη ενεργειακή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σε πολιτικό επίπεδο. Ε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, βεβαίως ε, η φτηνή ενέργεια είναι σημαντική. Η αλλαγή ε, από τις παραδοσιακές κεντρικές μονάδες παραγωγής της αποκεντρωμένες είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέους συμμετέχοντες στην αγορά και να βασίζεται η ενέργεια σε ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει να πιέσουμε για ένα μοντέλο που ενισχύει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μόνο δικός μου στόχος, αλλά έχει οριστεί και από τον Γιούνκερ, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να είναι η παγκόσμια πρώτη ένωση, ε, ε, αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε πρέπει να διατηρήσουμε τη στάση αυτή. Για τον κανονισμό τώρα για το σχεδιασμό της αγοράς θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σωστό, ωφέλιμο πλαίσιο για νέους συμμετέχοντες, για τα προγράμματα στήριξης και επίσης θα πρέπει όλα όλοι οι πολίτες να έχουν δικαιώματα και να μπορούν να επωφεληθούν από την ενεργειακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει αυτοπαραγωγή, καλύτερη σύνδεσμη με τις πόλεις ε, ε, πώλησης αγορές και επίσης ενίσχυση συγκρισιμότητας των ε, ενεργειακών συμβάσεων. Και επίσης πρέπει να έχουμε ε, τάξεις που θα προστατεύουν τους πιο ευαίσθητους ευάλωτους ε, πολίτες μας. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνοχή, την τονίζω και υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, επιλεξιμότητα των μηχανισμών δυνατοτήτων που ερέ, με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για τον άνθρακα. Δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα πιο, α, τις μονάδες παραγωγής που, που παράγουν ενέργεια μέσω άνθρακα όταν υπάρχουν πιο καθαρές δυνατότητε παραγωγή ενέργεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Τερέζα. Ο κύριος Λόπες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένας νέος σχεδιασμός της αγοράς είναι απαραίτητος ε, ώστε να καλυφθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, αυτό χρειάζεται ρύθμιση για τις τιμές μέσω και ε, μακροπρόθεσμα και είναι απαραίτητες επενδύσεις για την καθαρή ενέργεια. Ωστόσο υπάρχουν αντιφατικές προτάσεις μέτρων οι μηχανισμοί αμοιβή ε, για τις, ε, την παραγωγική ικανότητα ε, θα πρέπει να δούμε, να, μην, να φροντίσουμε μάλλον να μην συνεχίζεται η παραγωγή ηλεκτρισμού από ρηπαίνουσες πηγές. Αντίθετα θα πρέπει να ευρωηθούν οι ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ξέρουμε ότι ακόμα δεν αρκεί, αλλά αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να συνεχίσουμε να παράγουμε ρηπαίνοντας. Ε, είναι καλή η πρωτοβουλία για να μπορέσει ο, ο πολίτης να ε, χειραφετηθεί στην ε, παραγωγή της δικής του ενέργειας μέτρα για να βελτιωθεί το ηλεκτρικό σύστημα και να αυξηθεί η συμμετοχή των καταναλωτών και ε, προσφέρω τη συνεργασία μου ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συνεμείς οι προτάσεις μας. Γιατί είμαι και εγώ εισηγητής για ένα άλλο κομμάτι της δέσμης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν τρία βασικά θέματα. Η τιμή, η ασφάλεια και το περιβάλλον. Και βεβαίως η μόλυνση και η κλιματική αλλαγή. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν για την ε, ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Πρέπει να τονίσουμε το θέμα των ε, κλιματικών αλλαγών. Έχουμε την Συμφωνία του Παρισιού και πρέπει να την τηρήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλές νέες τεχνολογικές λύσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, περισσότερες από αυτές που ακούστηκαν σήμερα. Ήδη υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στο στόχο μας αλλά πρέπει, έχουμε και, την, ε, και κάποιες ε, παραδόσεις οι οποίες ε, υποστηρίζουν τα λάθος εργαλεία και δυσκολεύουν τις υπάρχουσες δομές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε σε μεγαλύτερο εύρος και με καινούριο τρόπο για να μπορέσουμε να, να έχουμε λειτουργούσες αγορές. Να μην κοιτούμε μόνο τις υπάρχουσες δομές, αλλά και τις νέες δυνατότητες, τις νέες τεχνολογίες. Γιατί λοιπόν υποστηρίζουμε κάποιον από την ενεργειακή φτώχεια που ε, μπορεί να προωθήσει την ε, παλιά παραγωγή ενέργειας ε, που, είναι, που ρηπαίνει και δεν είναι καθαρή ενώ μπορούμε να έχουμε καλύτερες πηγές παρόλο που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβές. Οπότε ας δούμε τους, έχουμε ένα ρεαλιστικό τρόπο για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και ας δούμε τις ε, ευκαιρίες που έχουμε για να αλλάξουμε το σύστημα. Αλλάζουμε λοιπόν την παραγωγή, αλλάζουμε το σύστημα διανομής και έχουμε και για τα δύο πολύ με καινούργιες ε, τεχνολογίες ε, και φρέσκες λύσεις για να το κάνουμε. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε και να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία για να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα να δούμε τις ε, διασυνδέσεις, τους κανόνες που υπάρχουν, οι οποίοι επίσης είναι ε, ανθρωπογενείς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο... να έχουμε καλύτερο όραμα για αυτές τις ε, νέες αλλαγές που θέλουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ζωχίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να κάνω τη συμβολή μου σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Η ενεργειακή μετάβαση σημαίνει ότι πρέπει, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε από πού ξεκινάμε, αλλά κυρίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα από του λίγου τομεί όπου η Ευρώπη θέλει και μπορεί να ηγηθεί. Επίση, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε και να λάβουμε υπόψη την ποιότητα ζωή και την ποιότητα του περιβάλλοντο. Αυτή η ενεργειακή λοιπόν ε, ηγεσία δεν θα πρέπει να θέσει ένα αμφιβόλο την ε, κατάσταση των επιχειρήσεων ούτε και των πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σταδιακή πορεία, να φτάσουμε να έχουμε μια ένα αποθεματικό που μπορεί να είναι πυρηνικό, που εγώ δεν είμαι υπέρ, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχει ήδη, μπορεί να είναι εκεί το αποθεματικό, μπορεί να είναι συνδυασμένο αποθεματικό, μπορεί να είναι τα συστήματα ε, ε, νερό, αέρας, ε, ήλιος και έπειτα η αγορά θα εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε δίκτυα ολοκληρωμένα ενέργειας που η συνεργασία είναι θεμελιώδης και κάθε φορά θα έχουμε αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση σε μικροσυστήματα οπότε ο συντονισμός της απόδοσης είναι καθοριστικός. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μικροδιάσταση και την ε, μακροδιάσταση. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το σχήμα, τη μορφή της διακυβέρνησης της Ενεργειακής ε, Ένωσης. Όλα θα συνδέονται με όλα ε, και γι' αυτό καλό τους συναδέλφους να κάνουμε μία προσπάθεια κοινού στρατηγικού οράματος ολοκλήρωσης ακριβώς μέσα σε αυτό το σχήμα της διακυβέρνησης γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Αυτό που ήδη δεν λειτουργεί δεν θα λειτουργήσει ούτε στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Συνάδελφε Κάριν, σε πολλές προσδοκίες Α, συγγνώμη, ο κύριος Κόχλιτσεκ, δε, συγγνώμη, δεν σας είχα στον καταλογό μου. Μπορείτε να πάρετε το λόγο τώρα, ναι. θέλω να κάνω κάποιες πρακτικές φύσης παρατηρήσεις. Πρώτον, νέα ε, ενεργειακή αγορά και καταναλωτές δεν θα πρέπει αυτό να βαραίνει τους παραδοσιακούς καταναλωτούς. Κάθε φορέας θα πρέπει να φέρει το κόστος του ανάλογα με την συμμετοχή του στο ηλεκτρικό σύστημα. Στην περίπτωση του ομαδοποιητή αυτό σημαίνει τιμολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος της περιφερειακής ε, διανομής. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, ε, τους λεπτομερούς λογαριασμούς ενέργειας. Υπάρχουν τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Πολλοί καταναλωτές εξάλλου σήμερα διαμαρτύρονται για την περιπλοκότητα και την έλλειψη σαφήνειας στους λογαριασμούς. Έχετε δει τελευταία πώς έχουν οι λογαριασμοί. Είναι καταστροφή. Εγώ που είμαι τεχνικός, παρά το γεγονός ότι παράγω και ενέργεια, έχω πρόβλημα να καταλάβω το λογαριασμό. Πρόσφατα μιλούσαμε για την πρόσφατη αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού χωρίς λόγο, χωρίς κάποιο σαφή λόγο οι φορεί ε, διαχείρισης των συστημάτων διανομής θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία για να εισάχουν την ευελιξία στα δίκτυά τους με τον πιο ε, προσιτό τρόπο. Είτε πρόκειται για την αγορά είτε για, για αυτοδιαχείριση ώστε να επιβαρυνθεί όσο γίνεται λιγότερο καταναλωτή κάθε φορά. Και έπειτα η, η, η ευθύνη για την παροχή ηλεκτρισμού θα πρέπει να βαραίνει τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της διανομής. Η ευρωπαϊκή εναρμόνιση δεν θα είναι αποτελεσματική αυτή τη στιγμή. Και τελευταία παρατήρηση. Στην Γερμανία η γερμανική αγορά δεν υπάρχει. Σε μεγάλες χώρες Ήδη υπάρχουν περιφερειακές μόνο αγορές. Και, για και μόνο η υπερπαραγωγικότητα, η πλεονάζω παραγωγή μπορεί να δοθεί σε άλλα μικρότερα κρατημέλη. Ε, στο μέλλον θα πρέπει να αποφύγουμε αυτήν την ευθύνη γιατί μπορεί αυτό να ε, στρεβλώσει το σύστημα και να έρθουμε πάλι να βρεθούμε στο 19ο αιώνα όταν ε, εφευρέθηκε ο ηλεκτρισμός. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Το είπανε κάποιοι συνάδελφοι. 550 είναι το όριο για την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε το άρθρο 194, το ενεργειακό μείγμα, που είναι απόφαση του κάθε κράτους μέλους. Αν το κράτος μέλος θέλει να προωθήσει την ε, ε, επάρκεια μέχρι 40% και τις ε, ε, ανανεώσιμες ε, μέχρι το 50% και να μειώσει τον, ε, το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να το ορίσει το κράτος μέλος. Και να μην λέμε ευρωπαϊκά ότι είναι 550 το όριο. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Δεν έχω κανέναν άλλο να ζητάει το λόγο. Ξέρω ότι είναι συνεχής αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή μας, αλλά κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν και Ήθελα να το επαναλάβω. Μπορούμε να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, αν θέλετε, γιατί ούτως ή άλλω δεν είναι η αλλω δεν ειναι η τελευταια μας αφορά που συζητούμε το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό, για τις επενδύσεις, αλλά όχι για τις, για τις δυνατότητες, αλλά για τα δίκτυα, επενδύσεις στα δίκτυα. Γιατί στην περίπτωση της ε, διανομής, συνήθως υπάρχουν κρατικές εταιρείε. Αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας στην ενεργειακή αγορά από μεγάλες οντότητες, άνθρακα κτλ., ε, ε, εγκαταστάσεις παραγωγής, σε πιο... Ε, ε σε περισσότερες δυνατότητες αυτάρκειας. Βεβαίως το κόστος είναι μεγάλο και στα δύο, και στην διανομή και στην ε, μεταφορά. Οπότε το θέμα πάντα είναι το θέμα της, ε, των επενδύσεων και του κόστους. Αλλά για το δίκτυο έχουμε δύο θέματα. Καταρχάς έχουμε το ICT. Έχει προσθεθεί στις υπάρχουσες, ε, στα υπάρχοντα δίκτυα. Διανομής και μεταφοράς. Έχει γίνει αυτή η προσθήκη των ε, ευθείων δεκτήων Και επίσης κάτι άλλο που είναι τελείως καινούριο. Οι ε, γραμμές μεταφοράς. Εκεί έχουμε δύο τελείως διαφορετικά θέματα να δούμε. Για την ε, διανομή είναι πιο εμπορικό το θέμα, αλλά καταλαβαίνω ότι το τελικό κόστος βεβαίως θα το επομιστεί ο καταναλωτής. Αλλά στην αρχή της όλης διαδικασίας κάποιος πρέπει να καταβάλει τα χρήματα. Στο τέλος προφανώς το, τελικό κόστος θα το έχει ο καταναλωτής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Δύο ερωτήματα λοιπόν έχουμε να σκεφτούμε πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά την, τις επενδύσεις. Και τώρα, να ακούσουμε τον, ε, ε, τον ε, κύριο Μπόρχαρ, διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, να μας πει κάποια πράγματα για τα δύο αυτά νομικά κείμενα. Και σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα για να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω αυτή τη συζήτηση που κάνετε και βλέπω ότι οι δύο πράγματα είναι σαφή γενικώ και χαίρομαι. Με όλες τις αποχρώσεις που ακούσαμε, αυτό που βλέπω είναι ότι η Κομισιόν με την πρότασή της έχει θέσει το πλαίσιο για το μελλοντικό σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σωστά. Και οι στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε με το πακέτο αυτό είναι κοινοί. Τώρα, για τις λεπτομέρειες, και βεβαίω αυτό είναι φυσιολογικό. Προφανώς υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις για το πώς ε, θέλουμε να εκπονηθούν τα διάφορα στοιχεία της, πρόθεσης, της πρότασης. Τώρα, για τα όσα υπόθεκαν στη συζήτηση. Για το θέμα της, ε, του μηχανισμού του αντισταθμιστικού. Άκουσα την κυρία Νίμπλερ και συμφωνώ ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη ε, και εσείς ελπίζω κυρία Νίμπλερ, οι μηχανισμοί αντιστάθμισης θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι του συστήματός μας, αλλά θα πρέπει να είναι η τελευταία μας δυνατότητα. Το τελευταίο καταφύγιο, όχι το πρώτο. Πρώτα θα πρέπει να αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι καταλαβαίνει και η να προτείνει κάποια στοιχεία έτσι ώστε η αγορά να μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει τις νέες επενδύσεις, τις δυνατότητες ώστε να μην χρειάζονται αυτοί οι μηχανισμοί αντιστάθμισης, αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Αν το αποδεχτούμε θα πρέπει να είναι η τελευταία μας δυνατότητα και θα πρέπει η αναγκαιότητά του να αποδειχθεί σε περιφερειακή βάση και με βάση κοινέ μεθοδολογίες. Αυτό είναι σημαντικό. Ο πρόεδρος έδωσε το θέμα των 550 γραμμαρίων για το διοξείδιο του άνθρακα αυτή η απόδοση έχει και κάποιες, ε, έχει κάποια αιτιολόγηση. Δεν έχει καμία σχέση, κύριε Πρόεδρε, με το 194 που είπατε, γιατί δεν αποτρέπουμε την παραγωγή από άνθρακα. Αυτό που αποτρέπουμε είναι αυτή η παραγωγή να έχει πρόσβαση, όπως είπε και ένα συναδελφό σας, σε ε, επιδότηση τα περισσότερα προγράμματα μέχρι τώρα είναι προγράμματα επιδότησης. Και αυτό λέμε, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε νέες επιδοτήσεις για παραγωγή τέτοιου είδους. Και για τον κύριο Τσέσακ θέλω να πω ότι ανέφερε την ε, μακρόχρονη ανεξάρτητη παραγωγή. Ε, εδώ πάμε λίγο μακριά τώρα, γιατί αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, προμήθεια με φτηνό τρόπο, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να έχουμε υπόψη μας και τη διασυνοριακή πτυχή, το διασυνοριακό εμπόριο και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις εθνικές ε, ανεξάρτητες δυνατότητες παραγωγής. Τούτου λεφθέντος είμαι ο πρώτος που θα δεχτώ ότι κάθε κράτος μέλος από μόνο του μπορεί να χρησιμοποιήσει την εσωτερική του παραγωγή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι ο πρώτος του στόχος να φτάσει σε, πλή, σε 100% αυτάρκεια σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπε ο, κύριο, ο κύριος Τούρμας, και συμφωνώ, και νομίζω όλοι συμφωνούμε, η περιφερειακή συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε αν πιστεύουμε στο στο μέλλον της λειτουργίας της ιστορικής αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της περιφερειακής συνεργασίας πρώτα, η οποία θα ενισχυθεί μετά. Αλλά αν το πιστεύουμε αυτό, αν πιστεύουμε δηλαδή στην ε, περιφερειακή συνεργασία, αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και από κάποιε δομέ και από κάποιε αποφάσει. Όπω είπε και ο κύριο Τούρμε, δεν μπορεί να έχουμε διαιτησία σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν σε μια περιφερειακή αγορά στο εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται αυτή η δυνατότητα και νομίζω ότι η Κομισιόν εδώ έχει κάνει πολύ προσεκτικά την πρότασή της σχετικά για τις ζώνες τώρα των προσφορών. Εδώ νομίζω ότι πρέπει τα πράγματα να είναι σαφή. Αν θέλουμε να φύγουμε από το πρόγραμμα των επιδοτήσεων και να έχουμε μέσω της αγοράς επενδύσεις, οι αγορές θα πρέπει να έχουν σωστές ε, ε, δυνατότητες επένδυσης. Αν έχουμε συμφόρηση, θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και γι' αυτό έχουμε τις ζώνες αυτές προσφορών. Ε, τέθηκε το ερώτημα πώς μπορεί να αποφασίσει η Ευρώπη για, την ε, εσωτερική, για τις εσωτερικές ζώνες της Γερμανίας ας πούμε. Μα το θέμα δεν είναι η Γερμανία. Το θέμα δεν είναι να μοιράσουμε τη Γερμανία σε δύο ζώνες. Δεν ξέρω πώς θα, είναι, πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει με βάση ε, ανάλυση σωστή. Και Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριο Τούρμε. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερε αγορέ ε, ρευστότητα και θα πρέπει να έχουμε σωστέ τιμέ. Και θα, αυτό θα γίνει μόνο αν έχουμε σωστέ ζώνε προσφορών και τιμών. Μετά να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γκρίφιθ και την κυρία Βέρνερ που μίλησαν για πολύ σημαντικά θέματα όπως η ε, ενίσχυση, η χειραφέτηση των καταναλωτών και νομίζω ότι στις ε, μελλοντικές συζητήσεις μπορούμε να επικεντρωθούμε και σε κάποια επιμέρους στοιχεία, αλλά αυτό που απορρέει από τα σχόλιά σας είναι ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στη σκέψη μας και όταν έχετε ιδέες για την ε, ενίσχυση αυτών, εμείς ευχαριστώ να σας ακούσουμε, γιατί αυτή είναι πραγματικά τεράστια πρόκληση να έχουμε τους ε, ε, καταναλωτές ε, ενεργούς και συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης να διορθώσω κάποια πράγματα που ίσως να μην έχουν γίνει απολύτως κατανοητά. Καταρχάς για ότι δεν υπάρχει αυτό το grandfathering που λέμε. Όντω, το θέμα της, του priority dispatch έχει καταργηθεί και ισχύει μόνο για τις νέες εγκαταστάσει, όχι για τις υπάρχουσες. Και επίσης, οι νέοι κανόνες ε, των διαφόρων ε, ε, περικοπών βάζουν τις, τις ανανεώσιμες στο τέλος. Αν είναι δυσανάλογο το κόστος της συμβατικής ενέργειας, τότε πηγαίνουμε στις ανανεώσιμες, Αλλιώ όχι. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ήδη στην πρότασή μας, υπάρχει. Και για τον κύριο Νίκα, άκουσα το όσα είπατε, αλλά να σας θυμίσω την ε, κατάσταση στην Ρουμανία τον ε, Γενάρη. Είπατε ότι θέλετε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον άνθρακα όταν είναι χαμηλές οι ε, θερμοκρασίες κτλ. Να σα θυμίσω ότι τον Γενάρη οι θερμοκρασίε ήταν πολύ χαμηλέ στην Ρουμανία και δεν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον άνθρακα γιατί είχε παγώσει. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν να το χρησιμοποιήσετε και να τον... για να παράξετε ενέργεια, οπότε όλο το πακέτο δεν μιλά για την επιβολή στα κράτη-μέλη απόλυτη αλλαγή. Ε, δραστικής αλλαγής των συστημάτων τους. Απλώς θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Ένας από αυτούς είναι να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας σε ό,τι αφορά τους στόχους του, για, το, για το περιβάλλον και το κλίμα. Για τις ε, ε ταρίφες ε, κατανομής. και εδώ υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης σε ό,τι αφορά το πώς θα το εκφράσουμε γιατί θέλω να είμαι απόλυτα σαφής εδώ, δεν έχουμε πρόθεση να εναρμονίσουμε την, ε, ε, τους, τα τέλη διανομής. Θα είναι φιάλτης να γίνει κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολο δηλαδή, και επίσης εδώ έχουμε και το θέμα της επικουρικότητας. Και θα είναι αδύνατο να βρούμε εναρμονισμένο τρόπο για να το κάνουμε αυτό. Οπότε πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ε, δεν μιλάμε για εναρμόνιση, μιλάμε για περισσότερη ε, διαφάνεια. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να το υπολογίσουμε. Και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημά σας κύριε Πρόεδρε. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Ε, αποκεντρωμένη ε, ενεργο, ε, παραγωγή, καταναλωτές, επενδύσεις στα δίκτυα. Μιλήστε και για τα ICT. Και είναι απολύτω απαραίτητο. Αλλά δύο πράγματα εδώ. Όσο περισσότερο επενδύουμε στις έξυπνε ευφυεί τεχνολογίες, όσο επενδύουμε στην ψηφιοποίηση και στο ICT, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να διευρύνουμε και να ενισχύουμε τα δίκτυά μας, κυρίως ό,τι αφορά τη διανομή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τα πάντα και όλες τις ε, επενδύσεις. Ο μόνος λοιπόν τρόπος για να γίνει αυτός, κατά τη δική μου άποψη, είναι δύο. Έχει, είναι διτός. Πρέπει να περάσουμε από τα, από τα τέλη. Εδώ θέλουμε, χρειαζόμαστε τους εθνικού ρυθμιστές και επίσης οι ε, καταναλωτές ε, και η αποκεντρωμένη παραγωγή θα πρέπει να έχουν το δικό τους μερίδιο του κόστους του συστήματος. Όχι με βάση τη δυνατότητα, αυτό θα ήταν δυσανάλογο, αλλά ένα δίκιο μερίδιο. Και ακόμα στην πρόταση μας δεν το έχουμε λύσει αυτό. Είπαμε όμως ότι πρέπει να βρούμε έναν ανάλογο τρόπο, αναλογικό τρόπο να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι καταναλωτές που παράγουν ε, ενέργεια στα τέλη. Αυτό λοιπόν ακόμα παραμένει εκρεμές, αλλά πρέπει να γίνει και πρέπει να είναι δίκαιος ο τρόπος. Συνολικά λοιπόν πρέπει να πω ότι καλωσορίζω ε, το ότι έχετε πραγματικά στοχεύσει στα πιο σημαντικά σημεία της πρότασής μας. Εγώ βλέπω ότι στις συζητήσεις σας κινείστε προς μια πολύ καλή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά την πρότασή μας και βεβαίως ευχαρίστως να συζητήσουμε και άλλο και να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, να δούμε τα θέματα των τελών κτλ. Αυτά από εμένα και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ε, Απαντήσατε στα σχόλιά μου. Κάποια βεβαίως έμειναν αναπάντητα. Οπότε θα, θα πρέπει να μου απαντήσετε στο γιατί, επενδύουμε, γιατί επιδοτούμε το ένα και όχι το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε την ερώτηση αυτή να την απαντήσουμε αν είναι σε διμερές επίπεδο, γιατί πρέπει όντως να έχουμε σωστή διαχείριση όλων των πηγών. Κύριε ε, Κάρινς, έχετε 10 λεπτά μόλις. Γιατί στις 5 και 4 περιμένουμε τους συναδέλφους από τις γειτονικές χώρες της, Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θέλουμε να αρχίσουμε έγκαιρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω έξι σελίδες σημειώσεις. Θα είχα κι άλλες αν δεν μου έχει τελειώσει το χαρτί. Σημειώνω όλα όσα είπατε και βλέπω συνολικά κανείς δεν λέει ότι δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση, αυτή την πρόταση κανονισμού. Κανείς δεν λέει ότι ε, είναι λάθος ο τρόπος αυτός για να συνεχίσουμε. Αλλά συμφωνούμε όλοι ότι οι αγορές αλλάζουν. Η παραγωγή ενέργειας επίσης αλλάζει γίνεται πιο άτακτη σε κάποια, σε κάποια επίπεδα, γίνεται πιο αποκεντρωμένη. Οπότε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένας τρόπος για να προσαρμόσουμε την αγορά, έτσι ώστε να υπάρξει ασφάλεια για τις επενδύσεις στο μέλλον. Χρειάζεται αυτή η ε, βεβαιότητα. Αν μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε ένα σωστό κανονισμό, θα έρθουν και οι επενδύσει, θα, θα υπάρχει ανταγωνισμό, οι τιμέ θα είναι χαμηλέ όσο γίνεται και για να γίνει αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να, έχουμε, ε, να μειώσουμε στο δυνατόν περισσότερο τις, τις τη της αγοράς. Και οι στρεβλώσεις είναι ουσιαστικά οι επιδοτήσεις για οποιοδήποτε είδος ενέργειας, για την ε, είτε για την παραγωγή, είτε για την μεταφορά, για τη διανομή. Όλες οι επιδοτήσεις, κάθε είδος επιδότησης στρεβλώνει την αγορά. Το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί και αποτρέπονται οι επενδύσεις. Και μάλιστα καμιά φορά δημιουργεί και λάθος επενδύσεις. Οπότε το ερώτημα δεν είναι να επιτύχουμε το στόχο, γιατί το στόχο θέλουμε όλοι να τον επιτύχουμε, αλλά το θέμα είναι πόσο μακριά θέλουμε να φτάσουμε για να ορίσουμε τους όρους για την αγορά, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη σαφήνεια. Βεβαίως ο διάβολος πάντα βρίσκεται στις λεπτομέρειες και σίγουρα θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Προσβλέπω λοιπόν στην περαιτέρω συνεργασία μας και με τους σκιώδεις και με όλους όσους θα, θα υποβάλουν τροπολογίε. Θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά αυτή και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένο και πολύ αισιόδοξο γιατί είμαι απολύτω πεπισμένο ότι ο στόχο θα είναι σωστό. Πρέπει να έχουμε την αγορά, μια λειτουργούσα αγορά, πρέπει να έχουμε επενδύσει και είμαι σίγουρος ότι όταν ε, ε, μαζέψουμε τα μανίκια μας και βάλουμε το κεφαλικά το σίγουρα θα επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ συνάδελφε και για τα τελευταία σας σχόλια και για την περίληψη της συζήτησης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή που κάναμε. Λοιπόν, ε, η μελέτη της γνωμοδότησης θα γίνει στις 10 και 11 Ιουλίου 2017, ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Σεπτεμβρίου Οπότε έχουμε και κάποιες, ε, έχουμε τις, το, μεσημεριανό, το καλοκαιρινό συγγνώμη, διάλειμμα μεταξύ των δύο προθεσμιών. Ε, μελέτη των τροπολογιών 11-12 Οκτωβρίου και ψηφοφορία στην Ήτρα 28 Νοεμβρίου. Τα περισσότερα κομμάτια του πακέτου του, για την καθαρή ενέργεια θα, θα ψηφιστούν τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Σας απασχολεί βλέπω ο Κλοντ. Ελπίζω να μην σας ε, πείσει να ακολουθήσετε τις δικές του ιδέες, γιατί έχω κι εγώ τις δικές μου ιδέες να σας ενημερώσω. Είναι πολύ γρήγορος όμως. Είναι σπίτι Γκονζάλες ο Κλοντ. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην ανταλλαγή απόψεων με την ενεργειακή κοινότητα. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας συνάδελφοι από την ενεργειακή κοινότητα και τις συμβαλόμενες χώρες. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Είναι η πρώτη συνάντηση του, της, ολομέ, της κοινοβουλευτικής ολομέλειας της ενεργειακής κοινότητας. Θα ξεκινήσουμε στις 6.45 ε, και ελπίζουμε και ότι θα είναι πολύ καλή η συνεργασία μας με τον κύριο Γιάννου Σκόπατς, Διευθυντή της ε, Γενικής Γραμματείας της Ενεργικής Κοινότητας στη Βιέννη και να πω ότι πρέπει να σας ε, θυμίσω, συνάδελφοι της Επιτροπής Ήτρε, ότι η συζήτηση στην Επιτροπή μας έχει προγραμματιστεί ακριβώς λόγω αυτών των σημαντικών αλλαγών που υπάρχουν στη δική μας πολιτική για το πακέτο κλιματικής, ε, ε, καθαρής ενέργειας, συγγνώμη. Για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας και τις δραστηριότητές μας. Να σας θυμίσω ότι η ενεργειακή, η ε, ενεργειακή κοινότητα είναι διεθνής οργανισμός που συνδυάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, χώρες από την νότιο-ανατολική Ευρώπη και τη χώρα της Μαύρης Θάλασσας. Έχουμε έξι βαλκανικές χώρες, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία επίσης, που είναι όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν σε πολλές συζητήσει και κάποιους παρατηρητές επίσης, όπως την Τουρκία για παράδειγμα. Και να πω να εξηγήσω μάλλον ότι σήμερα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα εξή. Ε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ, Κλοντ Τούρμες και Νταν Νίκα, καθίστε κάτω. and Καθίστε όπου θέλετε, αλλά να μιλάτε πολύ πολύ σιγά. Δεν χρειάζεται να φύγετε. Μπορείτε να μείνετε. Okay, okay. Uh, uh, we need more quiet atmosphere. Λίγη ησυχία παρακαλώ στο ακροατήριο. Λοιπόν, για τη συζήτησή μας σήμερα. Ο Διευθυντής της Συνεργειακής ε, Κοινότητας θα κάνει μια εισαγωγή για την οργάνωση και την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα σε αφορά την εφαρμογή της, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την Ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό. Και η, ενεργειακή, ε, η σύμβαση της Ενεργειακής Κοινότητας βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Επίσης, ο κύριος Διευθυντής θα τονίσει τις απόψεις του για το ρόλο της ενεργειακής κοινότητας στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Και βεβαίως και για το, στο πακέτο για, την, για το αέριο. Γιατί η, το, για την ασφάλεια παροχής αερίου δεν, έχουμε, δεν την έχουμε στο, κομμάτι, στο πακέτο αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Ίσως να υπάρχουν να πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στη συνθήκη ε, για την ενεργειακή κοινότητα. Αν θέλετε να συμπράξετε μαζί μας. Και θέλουμε να έχουμε μια ενεργειακή κοινότητα όχι των 27 ή των 28, αλλά των 35, ή 36 ευρωπαϊκών χωρών. Είναι λοιπόν σημαντικό ίσως να, γίνουν κάποιες ε, αλλαγές. Κύριε Διευθυντά, αν μπορώ να σας ε, δώσω το λόγο για να ξεκινήσετε. Thanks lot, ε, Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τα μέρη που προέρχονται από τη Σερβία, Μαυροβούνιο, Κωσυφοπέδη, Ουκρανία, Βοσνία, Ερζαγοβίνη και όλου του υπόλοιπου τη ελληνική κοινότητα. Μιλούσατε για 8 συμβαλόμενα μέρη. Πρέπει να θα σα διορθώσω γιατί μόλι εχθέ το Γεωργιανό Κοινοβούλιο επικύρωσε το πρωτόκολλο προσχώρηση, οπότε τώρα είμαστε 8 τα συμβαλόμενα μέρη. <laughs> Yes, coming closer, but it's already there. Uh, energy community. Η ενεργειακή κοινότητα είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που βασίζεται στο κράτος ε, δικαίου. είναι και βασίζεται και στο κοινοτικό κεκτημένο, δεν βασίζεται μόνο στις νομοθεσίες του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ε, μπορείτε να δείτε το χάρτη που επεκτείνει την περιοχή ε, του κοινωτικού κεκτημένου πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ανέφερε ήδη ο καθηγητής Μπούζεκ, με Πορτοκαλί έχουμε και κάποιους παρατηρητές και τη Λευκορωσία ως υποψήφια χώρα για να γίνει παρατηρήτρια και ελπίζουμε θα γίνει μέλος της οικογένειάς μας σύντομα. Αφού είναι ε, Εφόσον μάλλον αυτή η ενεργειακή κοινότητα βασίζεται στο κάτω δικαίου και όχι σε ένα μνημόνιο συνεννόησης ή κάτι παρόμοιο, έχει παρόμοια δομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 το Δεκέμβριο όταν όρισε τι είναι Ενεργειακή Ένωση σχεδίασε και έναν ορισμό που λέει ότι η Ενεργειακή Ένωση σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση συν την ε, συνδελόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας χάρη σε την τροπολογία που υπέβαλε τότε ο καθηγητής Πούζετ για εκείνο το ψήφισμα. Είπα ότι βασίζεται στο κράτος δικαίου. Προσπαθεί να αντιγράψει πιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουμε πολύ πολύ παρόμοια δομή στους θεσμούς μας, δηλαδή ε, Ρυθμιστικό Συμβούλιο ε, που είναι το δικό μας άσερ, που μόλις το συζητήσατε στο ΙΒΕΣΜΕ για την καθαρή ενέργεια. Έχουμε ένα είδος core ε, ΠΕΡ που είναι το Permanent High Level Group. Έχουμε μια μίνι κομισιόν και έχουμε τα φόρα και έχουμε και την κοινοβουλευτική απαρτία που δεν είναι κοινοβούλιο, αλλά ελπίζουμε θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο και γι' αυτό και πρώτη φορά σήμερα ερχόμαστε επισήμω σε επαφή μαζί σα. Έχουμε ε, επίση παρόμοια διαδικασία ρύθμισης διαφορών, αλλά δεν έχουμε δικαστήριο. Το δικαστήριό μας είναι το, το Συμβούλιο των Υπουργών που ε, στο τέλος ε, καθο... αποφασίζει. Έχουμε και καλύπτουμε διάφορα θέματα, ηλεκτρισμό, εμπόριο, φυσικό αέριο, από θέματα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβάλλον, και ούτω καθεξής, ενέργεια, ε, και επάρκεια. Αλλά θα έλεγα ότι σιγά σιγά εκτό από ενεργειακή κοινότητα μετατρεπόμαστε και σε περιβαλλοντική κοινότητα. Θα θέλαμε αυτό να αποτελέσει λοιπόν μια πλατφόρμα για το πώς θα μπορέσουν να ε, ολοκληρωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν οργανισμό ο οποίος ε, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο περίπλοκο στοιχείο είναι το τρίτο ενεργειακό πακέτο και εδώ έχουμε μια σύντομη παρουσίαση όπου τα συμβαλόμενα μέρη μας τα βλέπετε. Βλέπετε σε ποιο σημείο βρίσκονται. Εκτός από την Βοσνία Ζεγοβίνη και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν ενσωματώσει τα πακέτα ίσως όχι απολύτως στην εφαρμογή, στην εκτέλεση, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ανέφερε και ο καθηγητή Πούζεκ, βρισκόμαστε και αντιμετωπίζουμε ένα δίλημα αυτή τη στιγμή, γιατί αναπτύσσουμε ένα κεκτημένο, το οποίο, όπω είπαμε, έχουμε αντιγράψει από την Ευρώπη, αλλά στα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών μελών υπάρχει ένα νομικό κενό. Αυτό το νομικό κενό πρέπει να το γεφυρώσουμε κάπως και γι' αυτό ακριβώς φέτος συζητάμε ε, πιθανές τροπολογίες στη συνθήκη όπου θα λέμε τα κράτη-μέλη της Ένωσης που συνορεύουν με την ενεργειακή κοινότητα που είναι 8 Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία θα σέβονται το ίδιο καθεστώς ε, όπως ε, και τα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά σημαίνει πως αυτοί τα συμβαλόμενα μέρη που θέλουν αυτό να ωφεληθούν θα πρέπει, οφείλουν να ενσωματωθούν ακόμη περισσότερο, δηλαδή να εξομοιωθούν ακόμη περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και προτείνουμε άμεση εφαρμοσιμότητα των κανονισμών που ισχύουν στην Ένωση, αρμοδιότητα ορισμένων ευρωπαϊκών θεσμών ε, και στην επικράτεια της ενεργειακής κοινότητας, ίσως να είναι αιρετική αυτή η ιδέα, αλλά το ΆΣΕΡ που ορίζει τη, ρυθμίζει την αγορά και τη διαφάνεια αυτή, θα μπορούσε να δεν ήταν ίσως τρελό να, και συγγνώμη για αυτήν την να φτιάξουμε ακόμα ένα άσερ στην ενεργειακή κοινότητα. Καλύτερα είναι το άσερ να ε, καλύπτει και τις δύο πλευρές. Να έχουμε καλύτερη επιβολή σε περίπτωση παραβίασης. Δεν έχουμε εμείς δικαστήριο όπως σας είπα, αλλά εσείς θα πρέπει να έχουμε καλύτερους μηχανισμούς επιβολής ε, της ε, σχετικής νομοθεσίας και στα θέματα επιδοτήσεων και ανταγωνισμού. Τι έχουμε τώρα επιτάπητος και προτείνουμε στα συμβαλόμενα μέρη μας. Η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη αυτό το υποστηρίζει. Ελπίζουμε και ότι το Συμβούλιο θα δώσει σχετική εντολή στην Κομισιόν, αλλά ε, μπορεί όλα μας τα συμβαλόμενα μέρη να μην είναι σε θέση να ε, πάρουν αυτό το πιο προοδευτικό τρένο και γι' αυτό έχουμε προετοιμάσει μια λύση για να διευκολύνουν μια συμμετρική συμμετοχή κάποιες χώρες να μείνουν σε αυτό το καθεστώς που είναι τώρα και κάποιες άλλες να προχωρήσουν περισσότερο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις. Η Ευρώπη δύο ταχυτήτων ίσως να δοκιμαστεί λοιπόν πρώτα στην ενεργειακή κοινότητα. Δέσμη για την καθαρή ενέργεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας τα συμβελόμενα μας μέρη με, μεταγράφουν πάντοτε τις ίδιες, ε, τα, τα ίδια κεκτημένο όπως στην Ένωση. Και γι' αυτό το καλούμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί νομίζω πως τελειώνει ο χρόνος μου. Ε, και θα σας δώσουμε, στείλουμε τις λεπτομέρειες γραπτός, ώστε να μην σας κουράσω τώρα με αυτές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αυτή ήταν η αρχική μου εισήγηση, αλλά νομίζω πως και οι βουλευτές μας αργότερα θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την, αυτή την σημερινή ευκαιρία. Ο πρόεδρος Μπούζεκ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, Γιάννης για την ε, τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τους συναδέλφους μας από τα συμβαλόμενα μέρη της Ενεργειακής Ένωσης από τα κοινοβούλια δηλαδή πρώτα τον πρόεδρο όλων των κοινοβουλευτικών εξ ονόματος Ενεργειακής Ένωσης τον κύριο Μοχάμετ Μουσταφά από το Κόσοβο. Έχετε τον λόγο κύριε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε Πούσεκ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην παρούσα συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να θέσουμε υπόψη σας τις απόψεις μας σχετικά με τις προκλήσεις που ε, αντιμετωπίσαμε για να ε, στήσουμε στα πόδια τους κάποιες πολιτικές για την καθαρή ενέργεια. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι επιτύχαμε πρόοδο στο τρίτο πακέτο και όπως είπε και ο κ. Σκόπατς έχει ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο για το τρίτο πακέτο σε όλες τις χώρες σχεδόν και στο Κόσοβο το οποίο Κόσοβο ε, είναι δεσμευμένο να συμμορφωθεί με το κεκτημένο για, την, ε, για τις οικοδομές, για τις πολιτικές, για τις στρατηγικές, για την εξασφάλιση της ενέργειας και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους λοιπούς καταναλωτές. Ο ρόλος της ενεργειακής κοινότητας είναι τεράστιος για να υποστηρίξει και να διασυνδεθεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις χώρες οι οποίες φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως βοηθήσει να συντιμηθούν οι χρόνοι ε, για ε, την προσέγγιση αυτή. Αλλά μην λησμονούμε ότι η αφετηρία για πολλές από τις χώρες μας είναι πολύ διαφορετικές. Οι αφετηρίες είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη ανανεώσιμες ενέργειες, ιδίως κάρβουνο και λιγνίτη, που επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν τέτοια προβλήματα και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας, με τα όργανά σας, για να απαλληφθούν οι επιπτώσεις αυτών των πηγών ενέργειας. Και ένα από τα σημαντικά προβλήματα για την περαιτέρω, τις περαιτέρω υποδομές είναι και η ανάγκη να γίνουν αναλύσεις κόστους ωφέλειας που θα συμβάλλουν στο να μειωθούν οι επιπτώσεις διότι ακόμα ε, τα ευεργετήματα δεν έχουν φτάσει μέχρι ε, τις κοινωνίες. Αυτό είναι ε, αντιληπτό πλέον και μεταξύ των επενδυτών αλλά και μεταξύ των θεσμών. Στο Κόσοβο αρχίζει και ισχύει νέα νομοθεσία για την εξόριξη και ορισμένα από τα ωφελήματα θα καταλήγουν, από τα κέρδη δηλαδή των δραστηριοτήτων αυτών, θα καταλήγουν στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες ε, έτσι θα μπορέσουν ε, να ε, θα τις ενισχύσουν δηλαδή στο να ξεπεράσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των τεχνολογιών αυτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Πρόεδρος Μπούσεκ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ομιλείται μονάχα εξ ονόματος της Βουλής του Κόσοβου, αλλά και εξ ονόματος όλων των κοινοβουλευτικών ανδρών από τα συμβαλόμενα μέρη, από τις συμβαλόμενες χώρες της ενεργειακής κοινότητας. Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. πολύ ενθαρρυντικές οι παρατηρήσεις σα αυτές για μα, διότι ε, πρέπει να κατανοήσουμε και ποια προβλήματα σα απασχολούν. Πρόκειται για αμοιβαία υποφελή κατάσταση και για τις δύο πλευρέ και για τα συμβαλόμενα μέρη και για τις χώρε μέλη τη Ένωση. Θα παρακαλέσω τώρα να λάβει το λόγο άλλο μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως, ο κύριος Πιτλισέτσκι που εκπροσωπεί την Βουλή της Ουκρανίας. Έχετε το λόγο κύριε. Ε, λέγομαι Πιτλισέτσκι, ο Κρανός και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας. Επιτύχαμε με την υιοθέτηση του τρίτου πακέτου ενέργειας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το περάσαμε λοιπόν στο Ουκρανικό Δίκαιο. Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας που ήταν πολύ σημαντική για μας, για την Ουκρανία, που μας φέρνει κοντύτερα στην Ευρώπη, διότι εμείς συναισθανόμεθα ως μέρος της Ευρώπης. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί σε κάθε σφαίρα των δραστηριοτήτων μας. Στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και για ολόκληρη την Ουκρανία αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου τα ευρωπαϊκά ιδρώδη μας ε, εμπνέουν και μας και θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα είναι σημαντικό για μας να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις αγορές. Και η δυνατότητα εμπορικών ανταλλαγών είτε στο φυσικό αέριο είτε στο ηλεκτρικό ρεύμα έτσι ώστε να συναποτελέσουμε και εμείς μέρο μιας μεγάλης αγοράς, ώστε οι παραγωγοί της Ουκρανίας, για παράδειγμα, να μπορούν να πολλούν ενεργεία στη Γερμανία, για παράδειγμα, στην Ισπανία. Για μας είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια παροχής ενέργειας. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο χρειάζεται και η Ευρώπη. Η δημιουργία λοιπόν των διασυνδέσεων και εγκαταστάσεων back-to-back για την μετάδοση της ενεργειάς είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Νομίζω και ελπίζω ότι θα μπορούμε να παίξουμε ως μία ομάδα Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και με τους συναδέλφους των άλλων γειτονικών χωρών στοχεύοντας στην ασφάλεια της παροχής ενέργειας στην περιοχή μας που είναι πολύ σημαντικό για όλη μας την ομάδα. Έτσι λοιπόν οι διαμεθοριακές ροές ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν το βασικό στόχο της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Μπούσεκ. Και τώρα, παρακαλώ, ο κύριος Μπεσίμ Μπεγκάη που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο του Κόσοβου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Γραμματεία της Επιτροπής Ενεργειάς σας που μας δίνει να έρθουμε να μιλήσουμε και να μεταφέρουμε την εμπειρία από τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλήσαμε για την μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό μας δίκαιο. Επ' αυτού εργαζόμεθα ως χώρα. Καμιά φορά πρέπει να εξασφαλίσουμε ωστόσο όχι μόνο τη μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο και τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στις χώρες μας, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που είναι αναγκαία στην περιοχή μας, έτσι ώστε το δίκαιο που δημιουργούμε να είναι λειτουργικό. Αυτό συμβαίνει στην περιοχή μας. Στο Κόσοβο έχουμε εγκρίνει τώρα το τρίτο πακέτο, υπάρχει και σχετική νομοθεσία. Άρα περάσαμε από την φάση της συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τώρα έρχεται η φάση της εφαρμογής και είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Δηλαδή κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι η περιφερειακή ροή της ενέργειας. Κόσοβο και Αλβανία που υποστηρίζονται από τη Γερμανία και με τους προπολογισμού μας Φτιάξαμε και γραμμή μετάδοσης 100 κιλοβάτ μεταξύ Κωσόβου και Αλβανίας, ε, Αλβανίας γιατί θέλουμε να υπάρχει λειτουργική ροή, αλλά δεν λειτουργεί, διότι δεν υπάρχει συνεργασία λόγω των κολλημάτων. Διότι η συμμετοχή του Κωσόβου τελούσε υπό την αίρεση της εγγραφής ε, της σερβικής εταιρείας στο Κόσοβο, που όμως δεν έχει εφαρμοστεί και αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλους μας. Εκατομμύρια λοιπόν που έχουν, μπει, έχουν ε, φτάσει σε επενδύσεις και όμως η ροή της ενέργειας δεν έχει εξασφαλιστεί, δεν είναι ελεύθερη και αυτό το πληρώνουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μας. Με την έννοια αυτή απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξετε. Γνωρίζω ότι δεν είναι άμεσης αρμοδιότητά σας να υποστηρίξετε ώστε η συμμετοχή μας να μην είναι πάντοτε με όρους και αιρέσεις. Ο κ. Κόπατς μίλησε για τις επιλύσεις διαφορών όπου μόνο το Συμβούλιο Υπουργών άρα μπορεί να κάνει, αλλά ούτε και αυτό είναι νομικά δεσμευτικό. Έτσι το μέλλον, όταν μιλούμε για τροποποιήσεις της ε, ενεργειακής συνθήκης, θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της επίλυσης διαφορών μεταξύ μελών. Διότι όταν βλέπουμε ότι ένα μέλος δεν σέβεται τη συνθήκη και βλάπτει τα συμφέροντα ολόκληρης περιφέρειας, όχι μόνο μιας χώρας, θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Το άλλο θέμα για μας είναι το project TAP με τον αγωγό φυσικού αερίου. Χαιρόμαστε για τις επενδύσεις που γίνονται στην Αλβανία. Ως Κόσοβο, ωστόσο, δείξαμε την διάθεσή μας να συμμετάσχουμε, διότι μιλούμε για το 2030, 2040, η 50. Πρέπει να είμαστε διασυνδεδεμένοι και να έχουμε κάποιες εναλλακτικές επιλογές για την παροχή ενέργειας. Ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μας δίνετε να είμαστε ενώπιον σας σήμερα για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την περιφέρειά μας. Ευχαριστώ, Πούζεκ. μεγάλη χαρά και η δική μας που σας βλέπουμε εδώ και έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σας για όλα τα θέματα. Γιατί για μας η δραστηριότητά σας είναι πολύ σημαντική. Γιατί είσαστε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία μαζί σας είναι πολύ σημαντική. Και έτσι ο Ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω αν κάποιους άλλους από εσά, συνάδελφοι των συμβολωμένων μερών της κοινότητας ενέργειας, αν κάποιος θέλει να μιλήσει. Εκτός βέβαια από τους τρεις που ήδη τοποθετήθηκαν. Άλλος δεν ζητεί. Καλώς. Έρχομαι στα δικά μας μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Πρώτος ο κ. Τούρμες. Ευχαριστώ Ζέρζη, ευχαριστώ που οργανώσατε τη συνάντηση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι ανταλλαγές αυτές απόψεων μεταξύ ημών των Ευρωβουλευτών και ημών με ύψιλον των ε, βουλευτών των γειτονικών μας χωρών. Εάν κατανοώ σωστά, η ασφάλεια ενέργειας σημαίνει ασφάλεια επενδύσεων. Αυτό που έχει γίνει και λόγω των ανερχόμενων λαϊκιστικών κινημάτων στην Ευρώπη τελούμε υποπίεση να μην προχωρήσουμε σε ταχεία ένταξη όλων των χωρών σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις, διότι οι διεθνείς επενδυτές αμέσως φάνηκαν πολύ λιγότερο πρόθυμοι να επενδύσουν και σε τμήματα των χωρών σας. Χάρη και στην προσωπική δέσμευση του Ζέζι Μπούζεκ, ωστόσο, τουλάχιστον για την ενέργεια, και όσο δεν έχουμε πλήρη συμμετοχή σας, πλήρη ένταξη των χωρών σας, μπορούμε να προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη διαρθρωμένη συνεργασία να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι στέρεο και το οποίο θα μπορέσει πια με τη σειρά του να προσελκύσει τους επενδυτές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι ερωτήσεις που συζητούμε εδώ και ήρθατε να μας δείτε σε μια μέρα που συζητούμε τους νέους κανόνες και κανονισμούς και σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Αυτά καταστρώνουν το μέλλον της αγοράς ενέργειας. Ηλιακή, αιωλική, ανανεώσιμες και δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν. Αφενός ένα πολύ εύκαμπτο σύστημα, γιατί θα είναι διαφορετικές ανανεώσιμες ενέργειες από τις παραδοσιακές, και ένα ενδιαφέρον που έχουμε να ξεπεράσουμε τα σύνορα, δηλαδή να κάνουμε διαμεθοριακές κινήσεις. Αυτό που θεωρώ εγώ και είναι και ένα ερώτημα το οποίο συζητούμε εμείς εδώ οι ευρωβουλευτές, θέλουμε να επιταχύνουμε ένα είδος ρευστής αγοράς ενέργειας. Θα το κάνουμε αυτό μόνο για τις χώρες μέλη της Ένωσης ή θα πρέπει, και κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση, να φτιάξουμε ένα liquid power market, μια ρευστή ενεργειακή αγορά, και για τις χώρες μέλη αλλά και για τις γειτονικές αγορές για τις γειτονικέ χώρες, για την Νοτιοανατολική Ευρώπη ιδίως και ιδίως για την ηλεκτρική ενέργεια. Προσωπικά προτιμώ να συνεργαστούμε συλλογικά για να φτιάξουμε σταδιακά μια αγορά ενέργειας. Γνωρίζω για παράδειγμα ότι στη Σερβία δεν υπάρχει power exchange. Δεν είναι εύκολη η συζήτηση αυτή. Δεν μπορούμε, αν ο καθένα θέλει να παίζει πρωταρχικό ρόλο, να έχουμε 5 ε, ή 10 διαφορετικά χρηματιστήρια ενέργεια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μια περιοχή όπω η δική σα. Αλλά πού βρισκόμαστε, θεωρείτε ότι έχουμε συμφέρον να κινηθούμε ε, από κοινού προς την κατεύθυνση που περιέγραψα. Ένα άλλο θέμα είναι πρόσφατα στην διάσκεψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εναλλακτικών Ενεργειών που έχουν κάνει και μια μεγάλη μελέτη για τις ανανεώσιμες ενέργειες, το μήνυμα που δίνουν είναι ότι η περιφέρεια της Ευρώπης που έχουμε τις πιο φθηνές ανανεώσιμες ενέργειες δεν είναι οι χώρες του Βορρά, η Γερμανία, η Σουηδία κλπ. Ούτε καν η Πορτογαλία. Είναι η νοτιοανατολική Ευρώπη, διότι υπάρχει δυναμικό το οποίο δεν έχει ακόμα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε εκμεταλλευτεί όλο πλέον το υδροελεκτρικό δυναμικό μας, ενώ εσείς έχετε και πολύ ήλιο και πολύ αέρα. Άνεμο δηλαδή. Πού βρίσκεστε σε ό,τι αφορά την αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Ένα πρόβλημα που έχουμε δει στη Ρουμανία και Βουλγαρία για παράδειγμα, είναι ότι το κεφαλαιακό κόστος, το κόστος κεφαλαίου δηλαδή για τι ανεμογεννήτριες στην ε, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι στη Γερμανία για παράδειγμα. Τρία με 4% στη Γερμανία, 10 και 12% στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Αυτό που θέλουμε δηλαδή τώρα μαζί με τον κοινοτικό προπολογισμό, είναι να διατεθούν κίνητρα για να μπορέσει να μειωθεί το κεφάλαιο αυτό. η συμμετοχή δηλαδή του κεφαλαίου ως ποσοστό στην επένδυση. Άρα λοιπόν, αγορά ενέργειας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και το δεύτερο θέμα, το κόστος του κεφαλαίου για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ αγαπητέ Κλοντ. Κόχλιτσεκ με χαρά ακούω πολιτικούς που είναι τόσο καλοί και εξαίρετοι ρήτορες. Ε, δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι αλλού. Η νομοθεσία διέπεται από παραδοσιακή, ε, παραδοσιακή δομή στον τομέα του ηλεκτρισμού, όπου μετά τη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ευρωπαϊκά κράτη προσπάθησαν να ενοποιήσουν, να εναρμονίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές ε, στο χάλιβα, στον άνθρακα και είναι χαρά μας που σήμερα ακούμε ότι και τα γειτονικά μας κράτη θέλουν να σταθεροποιήσουν τεχνικά την κατάσταση, διότι όσοι έχουν εργαστεί στη βιομηχανία γνωρίζουν ότι μια γειτονική εταιρεία μπορεί να χαλάσει το δίκτυο εάν δεν ε, τηρεί τη εγκατάλληλη συχνότητα, βολτάζ κτλ. Και είναι χαρά μας να βλέπουμε ότι οι γειτονικές μας χώρες θέλουν να συνεργαστούν διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε διασυνδεδεμένα ε, ε, δίχτυα. Πριν 30-40 χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα ανάμεσα στην Ουγγαρία και την ε, Δυτική Ουκρανία που μπορούσαν να μεταφερθούν κάποια κομμάτια ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση και Τούμπαλιν και είναι χαρά μας να ακούμε σήμερα ότι μπορούμε να διευρύνουμε αυτές τις δυνατότητες. Βεβαίως, η σταθεροποίηση της συχνότητας, ε, του ε, εναλλασσόμενου ρεύματος κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα σκεφτούμε, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, για να μπορούμε, ας πούμε, να ανάψουμε το φως σε δύο-τρία σπίτια μόνο, γιατί η διασυνοριακή συνεργασία είναι ουσιαστική και είναι χαρά μας να ακούμε ότι ε, θέλουμε να λειτουργήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα προς το συμφέρον του καταναλωτή, όχι μόνο στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την τσεχική Επιτερία Τσέσ όμως η, και η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν κακές εμπειρίες, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τιμολόγηση στι τοπικέ αγορές πρέπει να ταιριάζει με τις δυνατότητες των καταναλωτών. Εγώ είμαι τεχνικός, δεν είμαι οικονομολόγος, οπότε καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από εκείνα τα μεγαλοαφεντικά που αγόρασαν κομμάτια των δικτύων και, κάποιες, και κάποια μεγάλα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγικά εκεί. Οι, τα, οι δεν είναι λύση σε όλα τα προβλήματα. Ε, υπάρχει πρόβλημα, για παράδειγμα, εδώ στις Βρυξέλλες, στην επίσκεψή σας, θα είδατε πέντε φορές να λάμπει λαμπρός ο ήλιος και πέντε φορές να βρέχει αν είχε όμως κανείς μια ε, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τον ήλιο, φανταστείτε τι σοκ έχει ε, κάθε φορά που πέφτει σε νεφιά. Το ίδιο και με την αιωλική ενέργεια γίνεται. Είμαι βέβαιος ότι θα χαλούσε τελείως το δίκτυο. Πρέπει πολύ προσεκτικά να εντάξουμε αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά την ε, δύναμη του νερού ή τη βιομάζα, εκεί είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί θα, μπορούσε ακόμα και να θα μπορούσαν ακόμα και να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση του δικτύου γιατί είναι πιο σταθερή η παραγωγή εκεί. είναι σοφό που δεν ακολουθείτε τυφλά οποιαδήποτε σύσταση. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε ότι είστε κομμάτια αυτής της κοινότητας. Αυτή η κοινότητα έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της και με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας στο μέλλον. Uh, <clears throat> uh thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κι εγώ κάποια σχόλια. Αναφέρατε το ενεργεια, την, δέσμη για την ενέργεια που εφαρμόζεται πλήρως ή σχεδόν πλήρως σε μερικές χώρες ε, που είναι συμβαλόμενα μέρη σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από άποψη επενδύσεων, όπως είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμβουλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας διότι χωρίς την εφαρμογή αυτού του σημαντικού πακέτου μέτρων δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως το τρίτο πακέτο για την ενέργεια. Επίσης, η δικτύωση είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε πλήρως να ανοίξουμε τα σύνορά μας για την ενέργεια. Έχω τρία ερωτήματα. Το θέμα αυτό που είπατε για το νομικό κενό στα σύνορά μας είναι σημαντικό να ε, καλυφθεί αυτό το κενό βέβαια. Και είπατε για αλλαγέ στη συνθήκη. μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι βέβαια η συνδραστηριότητα εντό του Άσερ θα είναι πλήρης και στην SOG και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ίσως μια τελευταία ερώτηση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Εάν θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά και να προχωρήσουμε σε επενδύσεις στις χώρες σας, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους παροχής για το φυσικό αέριο πούμε, από ορισμένες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό και σε επενδύσεις σε αυτή την περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες νομοθεσίες εφόσον υπάρχουν προβλήματα έρευνα κτλ. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατανοώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τη θέση σας γενικά, θα πρέπει να δούμε βήμα-βήμα πώς θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση. στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κάπως πιο εύκολη ολοκλήρωση, γιατί είναι σαφές ότι είναι προς το συμφέρον των συμπολιτών μας ε, ε, και το βλέπουν αυτό οι πολίτες. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει η γεωπολιτική, αλλά τους ενδιαφέρει να μην σταματάει η παροχή φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού Γι' αυτή την άποψη λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παροχή ηλεκτρισμού για τους πολίτες μας και εσείς θα μπορούσατε επίσης πολύ να βοηθήσετε και από την άποψη των ε, διάβλων προμήθειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, συνάδελφοι, να ρωτήσω αν έχετε κάτι να προσθέσετε εκπρόσωποι των συμβαλόμενων μερών μετά από τις δικές μας παρατηρήσεις Έχετε κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ. Ο συνάδελφος από την Ουκρανία, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Αναφέρατε τη γραμμή ηλεκτρικού που περνούσε από την Δυτική Ουκρανία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κομμάτι της Ουκρανίας είναι συνδεδεμένο ήδη με το πλέγμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ονομάζεται νησίδα Μπούστεν, τη γνωρίζετε φαντάζομαι, και ελπίζουμε στο μέλλον πως θα έχουμε ε, σύνδεση για ολόκληρη την Ουκρανία. Αν όχι τόσο γρήγορα, ε, πάντως θα μπορούσαμε να έχουμε δυνατότητες back-to-back για να μπορέσουμε να ε, εμπορευτούμε και θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει για κάποιες στιγμές στην Ευρώπη και κάποιες στιγμές και την Ουκρανία. Για μας αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτή η δυνατότητα back-to-back -back, ώστε οι τιμές στην χώρια αγορά είναι πολύ ψηλότερες στην Ουκρανία από ό,τι στην Ευρώπη <laughs> αυτή τη στιγμή για τον ηλεκτρισμό. Άρα λοιπόν θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει η Ευρώπη. Και για μας θα ήταν καλύτερο γιατί θα είχαμε χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή μας, αν μπορούσαμε να εισάγουμε ευρωπαϊκή ηλεκτρική ενέργεια. Καλή δυνατότητα λοιπόν για τις δύο πλευρές. Έχουμε πάνω από 40 εκατομμύρια κόσμο Μεγάλη χώρα είμαστε και γι' αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε αλλήλως. Και όταν μιλάμε για τον πράσινο τομέα, στην Ουκρανία έχουμε τις ψηλότερες τιμές για την ηλιακή και για την αιωλική ενέργεια. Έχουμε μεγάλη άνθηση στις επενδύσεις κατά συνέπεια. Και όπως είπε άλλος συνάδελφος, είναι πολύ καλός ο πράσινος τομέας, αλλά η εξισορρόπηση είναι πολύ σημαντική. έχουμε μια άλλη πρόταση για τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Έχουμε μια κρατική εταιρεία συν παραγωγής ηλεκτρισμού που έχει τρία μεγάλα εργοστάσια στην Ουκρανία και τώρα έχουμε πρόταση από Ευρωπαίο επενδυτή να το αγοράσει και να λειτουργήσει στην Ουκρανία. Έχουμε μεγάλη αγορά στην Ουκρανία με πολύ σπουδαίες δυνατότητες για το μέλλον. Τέτοιου είδους λοιπόν διασυνοριακή συνεργασία για μας είναι ζωτική σημασίας και νομίζω ότι έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλοί εταίροι, όπως είμαστε εδώ και χρόνια, στον τομέα του φυσικού αερίου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να παρέχουμε και ηλεκτρική ενέργεια και να είμαστε υπεύθυνοι εταίροι. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία σας και ελπίζουμε Πώ τέτοιε συνεδριάσεις θα γίνονται όλο και πιο συχνά και ευχαριστούμε και τη Γραμματεία που μα βοήθησε να φτιάξουμε τους κανόνες μας ε, όπως στην Ευρώπη. Γιατί άμα δεν έχουμε κοινέ νομοθεσίες δεν θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Η τεχνική συνεργασία είναι κάτι διαφορετικό από την νομική συνεργασία. Ε, πρέπει να έχουμε λοιπόν συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για να είναι αποτελεσματική. Έχουμε τώρα καλές δυνατότητες για επενδύσεις και είστε πρόσδεκτοι. Uh, uh, Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ουκρανία και στους αγωγούς αερίου επίσης είναι πολύ σημαντικές. Και για εμάς είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως πρέπει να προωθηθούν μέσω και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άλλος κανείς που να θέλει το λόγο, παρακαλώ από το κοσφοπέδιο. Ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις τους, τους ευρωβουλευτές. Έθεσαν και κάποια ερωτήματα. Για τις συμφωνίες ε, διανομής, έχουμε τέτοιου είδους ε, συμφωνίες. Δεν τις έχουν όλες οι χώρες στην περιοχή. Ας πούμε δεν έχουμε τέτοιου είδους συμφωνία με τη Φύρομ και με και διαπραγματευόμαστε τώρα μία με τη Σερβία. Οπότε αυτό είναι ούτως ή άλλως ε, εμπόδιο γιατί θέλαμε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις για να, να, να, αναβαθμίσουμε το δίκτυο διανομής που είναι σημαντικό για την ενεργειακή ροή. Οπότε έτσι δεν μπορούν να γίνουν ε, επενδύσεις ε, για μία μόνο χώρα γιατί τελειώς δεν έχει νόημα. Ως προς αυτό λοιπόν, δουλεύουμε σε δύο μέτωπα. Καταρχάς κάνουμε επενδύσεις που παίρνουν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν με την Αλβανία τουλάχιστον. Μιλάμε για 10 χρόνια να περάσουμε από την μελέτη σκοπιμότητα στην πραγματική αυτή καθ' αυτή επένδυση και εν τω μεταξύ προσπαθούμε να ε, απελευθερώσουμε και την αγορά. Παρόλο που έχουμε και ιδιωτική διανομή, Εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τι ιδιωτικοποίησει στο εσωτερικό τη χώρα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι εδώ δεν, δεν ιδιωτικοποιείται το δίκτυο. Η εταιρεία είναι ρυθμισμένη εταιρεία, είναι, ρυθμι, είναι ρυθμιζόμενες οι υποδομέ. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Και σε ό,τι αφορά το νομικό κενό, ναι, υπάρχει νομικό κενό. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε το νομικό κενό, υπάρχει εφαρμοστικό κενό της νομοθεσίας, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Ας πούμε, είμαστε στη διαδικασία να κατασκευάσουμε εδώ και 12 χρόνια μία εγκατάσταση. Εγώ ήμουν υπουργό Ενέργειας και η εμπειρία μου με την Παγκόσμια Τράπεζα και με, τα διεθνή, με όλους ήταν πραγματικά άσχημη. Και μάλιστα έλεγα στον Πρωθυπουργό μου, δεν θα τα καταφέρεις να φτιάξεις την εγκατάσταση αυτή με τις απαντήσεις που παίρνεις από τα θεσμικά αυτά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί γενικώ ε, υπήρχαν πολλές ε, αντιφάσεις. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε ε, να προωθήσουμε την, προ... την προμήθεια πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για τις ενεργειακές νοροές και την σταθερότητα στην περιοχή είναι αυτά τα κέντρα τα ενίδη χρηματιστηρίου ας πούμε ενέργειας. Θα είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί αυτό από την πλευρά του ε, ε Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκεί χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη και τις ιδέες σας. Η Γερμανία ήταν αρκετά ενεργή προς αυτό και τώρα πρέπει να δούμε μια καινούρια στρατηγική. Για να μπορούμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για να ενσωματωθεί και η ροή στο μέλλον, στο δίκτυο, σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δικές σας εμπειρίες στην αγορά του κουσουφοπεδίου όχι μόνο βέβαια στο κοσμοπεδίο αλλά και σε όλη την περιφέρεια, γιατί η ενεργειακή αγορά δεν είναι μια αγορά μια χώρα μόνο, αλλά η ε, στρατηγική θα πρέπει να εκπονηθεί για όλη την περιφέρεια και μετά να, συμπληρω... να είναι συμπληρωματική η πολιτική για την περιφέρεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι για το θέμα της νομικής βάσης. Οι δραστηριότητες σας στα ευρωπαϊκά, με τα ευρωπαϊκά ε, με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ε, αφορά στο δικό σας ενεργειακό και εκτιμένο. Οπότε ίσως να πρέπει να αλλάξει η συνθήκη σας έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε προσκοπτα και στον NSOE και στον NSOG και στον Acer. Ο κύριος Τούρμας έχει το λόγο για το θέμα του κόστους για τις ανανεώσιμες. Ήταν ακριβές οι ανανεώσιμες, αλλά δεν είναι ακριβές πια. Οπότε, αν δημιουργήσετε μια αν έχετε ένα συγκεκριμένο το... τέλος, πρέπει να το προσαρμόσετε με βάση και τις ε, τιμές οι οποίες ε, βαίνουν μειούμενες. Ε, μας, μας πήρε πολύ καιρό να κατεβάσουμε τις τιμές. Και αν οι επενδυτές μπορούν να, οι επενδυτές μπορούν να έχουν ένα τεράστιο περιφόριο ε, κέρδους, τότε και εσείς θα έχετε ένα, μια μεγάλη όθηση. Οπότε αν θέλετε να έχετε τέτοια συστήματα επιδοτήσεων ε, θα πρέπει να έχετε και μια ευελιξία. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποια σεμινάρια ή εργαστήρια για το πώς μπορούμε να ε, κάνουμε διαγωνισμούς, πώς οργανώνονται οι διαγωνισμοί για την αιωλική ενέργεια κτλ. Έτσι ώστε να έχετε περισσότερο ανταγωνισμό, για παράδειγμα, μεταξύ των επενδυτών και να έχετε χαμηλότερες τιμές. Τώρα, για τον άνθρακα, έχουμε την ίδια συζήτηση εδώ και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι στον ίδιο πλανήτη ζούμε. Έχουμε την Συμφωνία του Παρισιού αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει μέλλον για τον άνθρακα. Ακριβώς επειδή έχουμε έναν πλανήτη και δεν μπορούμε να κάψουμε άλλο κάρβουνο. Οπότε αυτό που είναι δύσκολο για τους επενδυτές είναι ότι αν εσείς ως χώρα δεν έχετε ε, μια στρατηγική 15-20 χρόνων ας πούμε, ε, ο επενδυτής, αν έχετε μια πολιτική μια τριετίας, ο επενδυτής είναι πολύ προσεκτικός και πολύ συντηρητικός στις επενδύσεις του. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το λύσουμε θεσμικά. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κρατημέλη σχεδιάζουμε τέτοια σχέδια για το 2030 για την ενεργειακή επάρκεια, διασυνδέσεις, κλιματική αλλαγή. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορέσουμε να ε, αυξήσουμε την ορατότητα για τους ιδιωτές επενδυτές. Γιατί αν ο ιδιώτης, ας πούμε, ξέρει ότι η Βουλγαρία θέλει να έχει τόση ηλιακή ενέργεια, τόση ηλιακή ενέργεια ε, και ολική για τα επόμενα 20 χρόνια, μπορεί να τον ενδιαφέρει και να εμπλακεί και να συμμετάσχει στην ε, βουλγαρική αγορά. Και αν γίνει ένας διαγωνισμός, να τον ενδιαφέρει να συμμετάσχει. Έχετε αρχίσει να συζητάτε στην ενεργειακή κοινότητα το θέμα αυτό. Δηλαδή θα μπορούσατε να προβλέψετε την επόμενη ε, δική σας, ε, το, τα επόμενα δικά σας βήματα με βάση και την μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί θα πρέπει να δώσουμε και στους επενδυτές ένα μήνυμα για το πού βρίσκονται οι αγορές σας και πού θέλετε να τις πάτε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Τούρμες. Θα ήταν ίσως καλό, ενθαρρυντικό για σας να μην συμφωνήσουμε για 100% για κάποια πράγματα. Όντως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε άνθρακα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καθόλου άνθρακα. Οπότε γενικώ θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η γενική προσέγγιση ωστόσο του Κλόντ είναι σωστή γιατί υπάρχει και η Συμφωνία του Παρισιού, είναι πολύ σημαντικό για μας να δούμε το μέλλον. Αλλά ας μην είμαστε πολύ γρήγοροι ως προς αυτό. Ας μην προτρέχουμε. Γιατί κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δυσκολευτούν. Δεν είναι ότι θα δυσκολευτείτε μόνο εσείς ως συμβαλόμενα μέρη. Ε, κάποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Το όνομά σα. Ο κύριος Φιλίπ Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Επιθυμώ να αρχίσω με την έκφραση της βαθύτατης ικανοποίησής μου όσον αφορά την συνεργασία με την Διεύθυνση Ενέργειας του κ. Γιάννη Σκόπατς. Βρίσκω ότι η συνεργασία αυτή κινείται προς τη κατεύθυνση για να επιλύσει βήμα-βήμα τα προβλήματα που διαπιστώνονται στον τομέα της ενέργειας και ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των χωρών της περιφερειάς μας, μεταξύ αυτών και η οικονομία του Μαυροβουνίου. Είμαι μηχανικός ορυχείων. Έχω και διδακτορικό ε, γεωλογίας. Έχουμε για πολλά χρόνια ε, προχωρήσει στην εξόριξη άνθρακα. Δεν θα σας μιλήσω τώρα όμως για το κάρβουνο για την ώρα το κάρβουνο ευθύνεται σε παγκόσμιο βαθμό για το 54% της ε, παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας. Δεν μπορεί να μείνει κανείς ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα της τάξης των 10-15 ετών θα μπορέσει να μειωθεί πολύ σημαντικά το υψηλό αυτό ποσοστό της συμμετοχής του άνθρακα. Όλοι οι ειδικοί ε, της ενέργειας το γνωρίζουν αυτό είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνει προσπάθεια για την μείωση της κατανάλωσης ε, άνθρακα. Αυτό μπορεί ίσως να γίνει μέσα στα πλαίσια μιας αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και στα πλαίσια της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που θα επιτρέπουν η υψηλότερη αποδοτικότητα. Με την επίτευξη υψηλότερων θερμοκρασιών από την καύση. Το Άνθακα για παράδειγμα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Όλες οι πηγές ανανεώσιμων ενεργειών από τη βιομάζα μέχρι την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια βεβαίως μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου αυτό είναι οικονομικά δυνατό. Για το Μαυροβούνιο έχουμε επιτύχει μάλιστα και τα ε, καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ενέργειες αυτές. Έχουμε βάλει ως στόχο ένα 30%, ένα κατόφλιο 30% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε ξεπεράσει το κατόφλιο μάλιστα αυτό και έχουμε φτάσει στο 40%. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το υψηλό αυτό ποσοστό συμμετοχής των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας του Μαυροβουνίου το Μαυροβούνιο ωστόσο είναι μια μικρή χώρα η οποία έχει και περιορισμένες ανάγκες σε ενέργεια και ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να εισάγουμε ενέργεια. Υπάρχει και η Ιταλική επιχείρηση η οποία πέρασε τα καλώδια της από το Μαυροβούνιο. Και υπάρχει και υποθαλάσσιο καλώδιο μάλιστα. Πολύ σημαντικό το καλώδιο αυτό για τη μεταφορά της στις ενέργεια από τα Βαλκάνια προς την Ιταλία. Η Ιταλία άλλωστε είναι ε, πολύ σημαντική χώρα μέλος και η γειτονά μα από την μεριά της Αδριατικής θάλασσας. Όπως είπα, χρειάζεται μείωση της συμμετοχής του άνθρακα για την μείωση και των ε, δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα ότι όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να έχουμε τους ίδιους στόχους όσον αφορά το περιβάλλον. Όσο δεν επιταχύνεται πάντως η πορεία της ένταξης των μικρών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβούμε ότι θα παραμείνουμε στο επίπεδο των επιθυμιών, των ευχολογίων. πρέπει να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάσει το μέλλον της. Ένας αριθμός μικρών χωρών μελών αποφάσισαν λοιπόν να φτιάξουν μια μικρή ένωση 100 εκατομμυρίων για να προχωρήσουμε σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Αλλά εμείς θέλουμε να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα θα γίνουμε ε, μέλος του ΝΑΤΟ. Ε, μιλώ για το Μαυροούνιο. Πολύ σύντομα. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να ενταχθούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τι παρατηρήσει σα. Δεν βλέπω άλλον να ζητεί το λόγο. Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν τον αγαπητό... Α, με συγχωρείτε. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακόμη παρούσα. Ο κύριος Ρόντερικ Βαν Βόλστ Ο κ. Κόπατ είναι μάλιστα και αυτό μέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίο εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Βιέννη. Μπορείτε λοιπόν εσεί υπάρχει εκπροσωπή τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κάνετε κάποια σχόλια. Έστω και αν τελικώ θεωρηθεί ότι πρόκειται για μια εσωτερική συζήτηση μεταξύ δύο συναδέλφων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τον ένα εννοώ τον κύριο Κόπατς. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά που μου δίνετε τη δυνατότητα να ομιλήσω. Δεν είμαστε ακριβώ συνάδελφοι ο Γιάννη Κόπα και εγώ. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Συμμετέχω και για θέματα διεύρυνση και ο κ. και η ομάδα του ε, είναι τοποθετημένοι αλλού. Ο κ. Κόπατς είπε στην αρχή της παρεμβάσεως του ότι η ε, γραμματεία της ε, κοινότητας ενέργειας είναι κάπως σαν την Κομισιόν. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι είναι. Αλλά λεπτομέρεια θα μου πείτε είναι αυτό. Θα είμαι σύντομο στην παρέμβασή μου. Θέλω να τονίσω ιδίω ότι η ανταλλαγή απόψεων που παρακολουθήσαμε μόλις δείχνει τις προκλήσεις αλλά και το πόσο σημαντικό είναι το έργο που κάνει η Γραμματεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι μιλούμε πρώτα για την εξασφάλιση του ότι οι συμβαλόμενες χώρες κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να αφομοιώσουν την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία. Είναι πολλή δουλειά αυτή. Ο δε πρόσωπος του Κωσόβου προ ολίγου αναφέρθηκε και στο κενό εφαρμογή το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην χώρα του για ορισμένα ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται η δουλειά για να εξασφαλιστεί ώστε το εφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο μεταφέρεται στα εθνικά δίκαια των συμβαλόμενων χωρών και εφαρμόζεται σωστά. Όπως είπα, αυτή είναι πολύ και βαριά δουλειά. Ένας αριθμός των συμβαρώμενων χωρών τα πάνε καλά, λίγο πολύ. Το Μαυροβούνιο, για παράδειγμα, είναι υπόδειγμα. Άλλες συμβαλόμενες χώρες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα για διάφορους λόγους. Είναι όμως μια προσπάθεια που συνεχίζεται και καταναλώνει και πολύ χρόνο και προσπάθεια καθημερινά. Δεν γίνεται πάντοτε με μεγάλη επιτυχία ή πάντως όχι έγκαιρα. Υπάρχει και μηχανισμός επιβολής στην βάση της συνθήκης και με τον οποίο προσπαθούμε να αναγκάσουμε των εισαγωγικών τι συμβαλόμενε χώρε να έρθουν στο ύψο των δεσμευσιών του. Γίνεται όπω είπα πολύ δουλειά. Ταυτόχρονα και είναι το δεύτερο που θέλω να τονίσω, ο Ευρωβουλευτής σας κύριος Τούρμες ζήτησε από τις συμβολόμενες χώρες να αρχίσουν να σχεδιάζουν ίδια το 2030. Έχει δίκιο που το κάνει αυτό, διότι με τον τρόπο αυτό παραπέμπει στο εργό το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται, που αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και συμβαλωμένων μερών από την άλλη σχετικά με το ποια ευρωπαϊκά νομοθετήματα ποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα συμβαλόμενα μέρη. Διότι δεν έχουν συμφωνηθεί όλα όσα θα ανατεθούν στις συμβαλόμενες χώρες. Υπάρχουν εκεί κάποια κενά. Ιδίω βεβαίω το πακέτο καθαρής ενέργειας προωθούμε με την έγκριση του πακέτου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν θα εγκριθεί, ή πάντως όταν θα εγκριθούν τμήματα του πακέτου αυτού, αυτό θα σημαίνει νέες προκλήσεις στο μέλλον για τα συμβαλόμενα μέρη. Ταυτόχρονα κοιτάζουμε προς το μέλλον μαζί με τα συμβαλόμενα, χώρα, ε, με τα συμβαλόμενα ε, μέρη. Και έρχομαι έτσι στο τελευταίο σχόλιο μου. Μέρος της εργασίας αυτής που είναι στραμμένη προς το μέλλον, ώστε να είναι έτοιμη για το μέλλον η κοινότητα ενέργειας, βασίζεται και στη συζήτηση δυνατοτήτων τροποποίησης της συνθήκης ενεργειακής κοινότητας για να είναι πλέον κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της δουλειάς μας την οποία βασίζουμε στην έκθεση που συντάχθηκε από την υψηλή ομάδα προβληματισμού της οποίας ηγηθήκατε εσείς κύριε καθηγητά και συχνά στην Επιτροπή μιλούμε για την έκθεση Μπούζεκ. Συνεργαζόμαστε με τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας για να επιφέρουμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας, ώστε να προσαρμοστεί αυτή καλύτερα στα μελλοντικά της καθήκοντα. Δεν θα αναφερθώ σε περισσότερα από τα στοιχεία που ανέφερε στην τοποθέτηση του Διευθυντής κ. Σκόπατς, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών του Οκτωβρίου θα μπορέσει να καταλήξει τουλάχιστον στην έγκριση ενδιάμεσων, προσωρινών πορισμάτων ή συμπερασμάτων. Ευχαριστούμε πάντως τα συμβαλώμενα μέρη για τη διάθεσή τους και τη συνεργασία τους μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μπούσεκ, για τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σας. Μιλήσατε για την έκθεση, ε, της οποίας υπήρξα, υπήρξα με άλλους. Εκεί προβλέπαμε τρεις, τρία επίπεδα βελτιώσεως. Πρώτα, στην βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων, για την εφαρμογή τους στο βαθμό που ήταν αναγκαίο. Δεύτερο, κατέστη αναγκαίο να ληφθεί απόφαση από τους Υπουργούς Ενέργειας, κάτι πιο περίπλοκο βέβαια, χωρίς αλλαγές στη συνθήκη. Και το τρίτο επίπεδο, πιο μακροπρόθεσμες προτάσεις και ευρύτερες προτάσεις για αλλαγές στη συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας. οι προτάσεις των δύο πρώτων επιπέδων εφαρμόστηκαν από τα συμβαλόμενα μέρη. Τώρα βρισκόμαστε στο επίπεδο 3. Τέλος πάντων αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα στην πρόταση αυτή. Και βέβαια αυτά ήταν και πριν από μια τριετία. Φίλε Γιάννη, κύριε Διευθυντά, εσείς. Uh, I would like to briefly answer, um... Ευχαριστώ πολύ να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Κλωτούρμες ανέφερε δύο πράγματα. Το ένα είναι εμπόριο τον, στον ηλεκτρισμό και το άλλο ήταν ανανεώσιμες. Όταν μιλήσατε για εμπόριο, Είπατε σωστά ότι δεν πρέπει να είναι μόνο περιφερειακό το εμπόριο, αλλά η ενεργειακή κοινότητα έτσι φτιάχτηκε για να οργανώσουμε το φερειακό εμπόριο. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται κανένα παράλληλο ω οργανισμός, θεσμός, οι νέες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε ήδη για την περιφερειακή συνεργασία. Λειτουργεί αρκετά καλά η δική μας κοινότητα. Εμείς ε, στην κοινότητα αυτή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα με τη σειρά από το περιφερειακό επίπεδο. Στο Πότκορη στο Μαυροβούνιο κατά κάποιο τρόπο επιβλήθηκε το να φτιαχτεί ένα γραφείο διαχείρισης των, ε, της παραγωγικής ε, λειτουργεί ικανοποιητικά παρά το ότι δεν συμμετέχουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν συμμετέχουν, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε. Πολύ καλύτερα, πολύ πιο εύκολο είναι να αναπτύσσονται ιδέες από κάτω προς τα πάνω, μην επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω. Και γι' αυτό εμείς ως γραμματεία δεν θέλαμε να φτιάξουμε ε, περιφερειακό και ανταλλαγή ε, ε, ηλεκτρισμού. Γιατί απλώς υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να το κάνουν. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ορισμένε χώρες ε, πριν από 15 χρόνια μόλις είχαν πόλεμο. Αλλά προσπαθούμε να αναπτύξουμε εθνικές ιδέες που σιγά σιγά θα πάρουν περιφερειακό χαρακτήρα. Όπως ε, το σερβικό χρηματιστήριο ενέργειας, που σιγά σιγά ε, προσελκύει φορείς από γειτονικές χώρες και το ίδιο έγινε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή υπήρχαν μόνο εθνικά χρηματιστήρια ε, ηλεκτρισμού και τώρα και σιγά σιγά προέκυψαν κάποια περιφερειακά και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να έρθουν σε διμερές ρίσεις επαφές και διμερές λύσεις με τις γειτονικές τους χώρες. Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να χρησιμεύσει ως ε, παράδειγμα σε αυτό το τομέα γιατί λειτουργεί πολύ καλά. Γιατί η πρώην Ιουγκοσλαβία λειτουργούσε πολύ καλά. μέσα. Όλοι μας, ε, όλα μας τα συμβαλόμενα μέρη, ε, κατά κάποιο τρόπο, εισήγαγαν τα ε, τέλη και ε, τα ρήφες για το ιδιωτική παραγωγής ρεύμα που μπαίνει στο δίκτυο. Και υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην τιμή της αγοράς, υπήρχαν και πρίμα για την τιμή παραγωγής, αλλά μόνο τρία κράτη-μέλη μέχρι στιγμής της Ένωσης ήδη το έχουν εφαρμόσει. Σε δικιά μας περίπτωση η Αλβανία ήδη ε, υιοθέτησε μια νέα νομοθεσία περί ανανεώσιμων που είναι στην ουσία γραφή της γερμανικής νομοθεσίας. Και τώρα η Γραμματεία προετοιμάζει παρόμοια νομικές λύσεις για όλα τα άλλα συμβαλόμενα μέρη. Θα τις προτείνουμε και ελπίζουμε ότι θα τις εγκρίνουν, θα τις υιοθετήσουν. Και αυτή η εξέλιξη στις ανανεώσιμες είναι πολύ ενθαρρυντική. Ο εκπρόσωπο του Μαυροβουνίου είπε ότι είμαστε τέσσερι ποσοστιαίε μονάδε πάνω από τον τελικό στόχο του 2020. Σχεδόν όλα τα συμβελόμενα μέρη είναι πάνω από τον στόχο. Μόνο τρία από τα οχτώ έχουν ακόμα προβλήματα, ε, αμφιβολίες για την πορεία τους. Όταν μιλάμε για τα χρηματιστήρια ε, και την ανταλλαγή μάλλον ε, ηλεκτρισμού, βελτιώνεται, αλλά χρειάζεται συνεργασία περιφερειακή και με τις χώρες της Ένωσης. Δεν θα πρέπει να παραμελούμε το τι συνέβη αυτό το φετινό χειμώνα, που δεν έγινε και πρώτη φορά η Βουλγαρία επέβαλε απαγόρευση στην εξαγωγή ηλεκτρισμού, πράγμα το οποίο ε, οδήγησε σε αύξηση ε, τιμών του ηλεκτρισμού στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία. Εμείς ως γραμματεία βεβαίως πήραμε διαμαρτυρίες από την πρώην Ιγκοσλοβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αρχίσαμε μια διαδικασία μαζί με την Κομισιόν και τώρα συζητάμε ε, με την, και με τη Βουλγαρία σε τριμερή διάλογο πώς θα εξασφαλίσουμε την μη επανάληψη της παρόμοιας κατάστασης. Αλλά και με την Ένωση χρειάζεται περιφερειακή συνεργασία. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα συμβαλόμενα μέρη της συνεργικής κοινότητας θα βλέπουμε σε ένα ξεχωριστό σύμπαν. Στην Νότια ανατολικη Ευρώπη αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο με τη Μολδαβία και την Ουκρανία που δεν είναι συγχρονισμένες εκτός από αυτό το μπούστεν, το, την νησίδα μπούστεν στην ε, βόρεια δυτική Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι αρκετά μεγάλη για να φτιάξει την δική της εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και με επιτυχία. Ε, και πράγματι βοηθούμε τη χώρα σε αυτό. Όμως αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι να μην συγχρονιστεί πολύ γρήγορα, γιατί τεχνικά δεν είναι δυνατόν με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά να επιβάλλει να φτιάξει back-to-back -back σταθμούς. δηλαδη να γίνεται τουλάχιστον μια μικρή ανταλλαγή ε, ηλεκτρισμού, να δημιουργηθεί πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και βέβαια περισσότερη ασφάλεια προσφορά στον τομέα του ηλεκτρισμού. Ο καθηγητής Μπούζεκ ανέφερε τρεις τομείς. Το νομικό κενό πρώτα. Εσείς οι προβουλευτές συζητήσατε την ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο και το σχετικό κανονισμό πρόσφατα. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το νομικό κενό με τη ρήτρα Σουιτσόν στο άρθρο 15 που δεν υποστηρίχθηκε όμως από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως εγώ γνωρίζω, είπε ναι, εντάξει μια τέτοια ρήτρα, αλλά όχι στον κανονισμό. Πρώτα πρέπει να προέλθει μέσω μιας διεθνής, να περιληφθεί σε μια διεθνή συμφωνία. Γι' αυτό τώρα συζητάμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το κενό και πώς θα επιβάλλουμε μια ρήτρα switch on στην συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας που είναι ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε πώς εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσατε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εντάξει, δεν το συγκρίνω, δεν είναι απόλυτο το ίδιο, αλλά κάποιες αλλαγές είναι τόσο ε, δύσκολες και ελπίζουμε πως τελικά θα ε, το επιτύχουμε φέτος. Τώρα, τα συστήματα μας ε, για τα Μπορεί κάνει να φανταστεί ότι λειτουργούν παρόμοια, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Έχουμε το ΆΣΕΡ που θα μπορούσε να επιτρέψει τη συμμετοχή εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, τέτοιων χωρών. Και ήδη η εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου προσεκλήθη να συμμετέχει, γιατί το Μαυροβούνιο ε, τηρεί πλήρως το τρίτο ενεργειακό πακέτο και αυτό ήταν προϋπόθεση. Ο Σέρβος ρυθμιστής το ζήτησε, αλλά η Σερβία δεν τηρεί πλήρω το τρίτο ενεργειακό πακέτο, οπότε δεν μπορεί ακόμα να συμμετέχει. Η ΕΝΣΟΗ έχει πλήρη μέλη από τα συμβαλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας. Η Αλβανία έγινε πλήρες μέλος μόλις τον περασμένο μήνα. Οι δύο χώρες που δεν, τρεις χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη είναι το Κωσυφοπαίδιο, η Ουκρανία και η Μολδόβα το κοσυβοπίδι μπορεί να μπει, αλλά υπάρχει βέτο από τον ε, χειριστή του συστήματος της Σερβίας και η Ουκρανία δεν μπορεί ακόμα να μπει γιατί δεν εφαρμόζει απόλυτα πλήρως το τρίτο πακέτο. Όμω η NSUG δεν δέχεται κανένα νέο μέλο που δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει να αλλάξει το, καταστατικό τους. Γιατί ας πούμε ο χειριστής της Ουκρανίας που είναι πολύ σημαντικός και πολύ αφοσιωμένος και που γνωρίζει και πάρα πολλά ασχολείται με, ως παρατηρητής με τις εργασίες της NSOG. Τελείωσα διαφορετική πολιτική. Ναι, ναι, ναι, κλείνω, κλείνω. επιβολή. Δεν μπορώ να πω πόσο πολύ συμφωνώ με αυτά. Ε, συμβαλόμενα μέρη μας... Ε, ε, αλλά βέβαια θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες. Εννοείται ότι χωρίς περαιτέρω νομική ολοκλήρωση αυτή η εσωτερική αγορά ενέργειας γιατί η ενεργειακή κοινότητα και τα μέλη της είναι κομμάτι της ενεργειακής αγοράς, δεν μπορούν να λειτουργήσει. Ε, και αυτό βλάπτει και ζημιώνει και την Ένωση. Εάν δεν λειτουργεί πλήρως η ενεργειακή αγορά στην Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει στον τομέα του φυσικού αερίου το ίδιο για την νοτιοανατολική Ευρώπη για τα θέματα ηλεκτρισμού. Οπότε δουλεύουμε πάνω σε όλα αυτά. Ε, αλλά νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά και σας ευχαριστώ για την τη σημερινή σας παρουσία εδώ και θα ε, ξαναπούμε σε 15 λεπτά στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Σαν θα συνεδριάσουμε ως Επιτροπή Ήτρε στις 20 ε, Μαΐου στο Στρασβούργο. 15. Μαΐου, μας συγχωρείτε, και 29 και 30 Μαΐου έχουμε πάλι νέα συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Ε, σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Πέρα τη σημερινή μας συνεδρίαση. αργήσαμε μόλις ένα λεπτό και οι διερμηνείς μας είναι ακόμα εδώ. Τους ευχαριστώ πολύ. Ε, σας εύχομαι ότι καλύτερο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στις Βρυξέλλες και σε 15 λεπτά εδώ ε, στην Κοινοβουλευτική συνέντευξη.